Gut, liebe Kolleginnen und Kollegen, dann setzen wir unsere Sitzung fort und kommen zu Punkt 9 unserer Tagesordnung. Και πάμε στο σημείο 9 της ημερήσιας διάταξης. Πρόκειται για το θέμα των προϊόντων καπνού και του εμπορίου αυτών στα πλαίσια του ΠΟΕ. Συγγνώμη, του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Θα δώσω το λόγο στον κύριο Σίνφελτ, τον ε, εισηγητή. Κύριε Πρόεδρε, πρόκειται για την πάταξη του παράνομου εμπορίου στα προϊόντα καπνού και τον έλεγχο αυτών των εμπορικών συναλλαγών. Πρόκειται ουσιαστικά για ένα πρωτόκολλο με πολύ μεγάλο τίτλο όπως βλέπετε, αλλά αυτή είναι η ουσία αυτής της ε, προσπάθειας. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει εδώ να δώσει τη συνένεσή του έτσι ώστε να ολοκληρωθεί αυτό το πρωτόκολλο. Για ποιο λόγο πρόκειται για την δραστηριότητα την οποία προσπαθούμε να ελέγξουμε. Πρόκειται για μια εγκληματική δραστηριότητα την οποία θέλουμε να πατάξουμε, δηλαδή την παράνομη παρασκευή, διάθεση στην αγορά, εμπορία, λαθρεμπορία προϊόντων καπνού. Και πέρα από το ότι πρόκειται για μια εγκληματική παράνομη δραστηριότητα, είναι πολύ σημαντικό να πούμε ότι φυσικά είναι κάτι που απειλεί την ζωή απειλεί την υγεία των Ευρωπαίων πολιτών. Και φυσικά αυτό μας προκαλεί και πολύ συγκεκριμένες οικονομικές ζημίες. Πρόκειται για μια παράνομη δραστηριότητα η οποία την ίδια ώρα ταυτόχρονα υπονομεύει και την αξιοπιστία των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όσον αφορά τις οικονομικές αυτές ε, απώλειες. Πρόκειται για 10 περίπου δισεκατομμύρια το χρόνο, άμεσες απώλειες, χωρίς βεβαίως ε, να υπολογίσουμε μέσα σε αυτό το ποσό και όλες τις ε, έμεσες οικονομικές συνέπειες που είναι η θεραπεία των ε, προκαλούμενων ασθενειών καθώς και όλες οι αγωγές για την απεξάρτηση αυτών των ανθρώπων που ε, είναι θυσμένοι στον καπνό. Ε, μιλάμε λοιπόν για παράνομη δραστηριότητα και για να είναι δεσμευτικό αυτό το πρωτόκολλο χρειαζόμαστε τουλάχιστον 40 μέρη στο πρωτόκολλο αυτό. Μέχρι τώρα έχουμε μόνο 15 κράτη-μέλη που έχουν ε, προσυπογράψει μάλλον που προτίθεται να προσυπογράψουν σημαντικά κράτη, Αυστρία, ε, Λετωνία, Ισπανία, Πορτογαλία. Πιστεύω ότι μόλις φτάσουμε τα 40 συμβαλόμενα μέρη, θα οδηγηθούμε και στην ε, πραγματική αποτελεσματική εφαρμογή των λύσεων που προτείνεται. Θέλουμε καταρχήν ένα σύστημα track and trace, ένα σύστημα το οποίο να παρακολουθεί όλη την αλυσίδα αυτών των προϊόντων καπνού αλλά και του εξοπλισμού και όταν αναφερόμαστε σε όλη αυτή την αλυσίδα βεβαίως αναφερόμαστε και στις άδειες, στην αδειοδότηση, στα Μητρώα, καθώς και σε όλες τις ρυθμίσεις που αφορούν τις εμπορικές συναλλαγές, την μεταφορά, το διεθνές εμπόριο. Δεν θέλω να μακρηγορήσω. Ξέρω ότι αυτό το πρωτόκολλο δεν έχει προκαλέσει πολύ σημαντικές αντιδράσεις. Προτείνω λοιπόν να το στηρίξουμε ε, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Καταρχήν θα ήθελα να ζητήσω συγγνώμη από τον Σέρτζο Γκουτέρες, ο οποίος ε, πρέπει να παρουσιάσει μια άλλη έκθεση στην ΙΜΚΟ αυτή την ώρα. Καλωσορίζουμε την πρωτοβουλία για τους ίδιους λόγους ε, με τον ε, συγγραφέα γιατί μιλάμε ιδιαίτερα για την παράνομη εμπορία προϊόντων καπνού. Πρόκειται για μια ε, παράνομη δραστηριότητα που υπόκειται σε ποινική δίωξη, δημιουργεί και προβλήματα υγείας, αλλά κυρίως γίνονται παράνομες εισαγωγές. Υπάρχουν στοιχεία που δείχνουν ότι μπορούν να χρηματοδοτηθούν και άλλες εγκληματικές δραστηριότητες όπως η τρομοκρατία. Το θέμα είναι πολύ σοβαρό. Όλα αυτά τα προϊόντα προέρχονται εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Χρειαζόμαστε διεθνή συνεργασία για να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση και το πρωτόκολλο προβλέπει τη διεθνή συνεργασία. Όπως είπε και ο εισηγητής, το πρωτόκολλο σχετίζεται με την αλυσίδα προμήθειας καθώς και τον τομέα της βιομηχανίας έτσι ώστε να υπάρχει ένα παγκόσμιο σύστημα ανείχνευσης και ιχνηλάτησης για να τηρούνται οι κανονισμοί, να υπάρχουν αφορολόγητα δίκτυα όπως τα duty free και άλλες αλυσίδες για να διατίθενται τα προϊόντα. Υποστηρίζουμε λοιπόν την κύρωση αυτή. Αλλά για να επικρίνουμε και κάτι, φαίνεται ότι απέχουμε πολύ η διεθνής διαδικασία είναι αργή. Ακούμε πολλά παράπονα για τη νομοθετική διαδικασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση που είναι πολύ αργή. Ε, υποστηρίζουμε όμως την κύρωση του πρωτοκόλλου. Ευχαριστώ. Έμα. Και... Και εγώ καλωσορίζω την πρόταση του συγητή να δώσουμε την συγκατάθεσή μας. Θεωρώ ότι το πρωτόκολλο αυτό δίνει μια λύση. Γνωρίζουμε ότι κάθε χρόνο 6 εκατομμύρια χάνουν τη ζωή τους από τις ασθένειες που προκαλούνται από τον καπνό και προβλέπεται αύξηση από τον ΠΟΗ. Γνωρίζουμε ότι ακόμα μεγαλύτερους κινδύνους εγκυμονούν τα προϊόντα τα παράνομα για την υγεία των ανθρώπων. Γι' αυτό θα έπρεπε η Ευρωπαϊκή Ένωση να ηγηθεί τις προσπάθειες που γίνεται να βρεθούν οι 40 χώρες που θα κυρώσουν το πρωτόκολλο αυτό για να τεθεί σε ισχύ. Χρειάζεται λοιπόν να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα αυτό που δεν είναι μόνο ευρωπαϊκό αλλά παγκόσμιο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Δεν ε, μπορούσε ο συνάδελφος να που είναι αρμόδιος για τους φιλελεύθερους να είναι εδώ σήμερα και αυτό μου ζήτησε να πάρω το λόγο. Στηρίζουμε πλήρως αυτό το πρωτόκολλο καθώς και την πάταξη του λαθρεμπορίου προϊόντων καπνού. Πρόκειται για μια εγκληματική δραστηριότητα με τεράστιες συνέπειες για την ε, δημόσια υγεία. Και βεβαίως ε, την ίδια ώρα πρόκειται για μια πηγή χρηματοδότησης ε, του οργανωμένου εγκλήματος, κάτι που δεν μπορούμε σε καμία περίπτωση να αφήσουμε να συμβαίνει. Όλα αυτά τα παραποιημένα και παράνομα προϊόντα συχνά προέρχονται εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης και βεβαίως χρειαζόμαστε και καλύτερη νομοθεσία και καλύτερη εφαρμογή της υπάρχουσας νομοθεσίας. Η φιλελεύθερη ομάδα πιστεύει ότι ένας τρόπος να πατάξει κανείς αυτές τις παράνομες διαδικασίες, την φοροαποφυγή, και φοροδιαφυγή, είναι να έχουμε καλύτερα ρυθμιστικά εργαλεία όπως ε, αυτή την συμφωνία πλαίσιο για τον έλεγχο των προϊόντων καπνού. Με μεγάλη χαρά λοιπόν θα ήμασταν υπέρ της ταχύτατης ε, υλοποίησης και εφαρμογή αυτού του πρωτοκόλου. Ευχαριστώ πολύ για την ΚΟΕ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πρόκειται για ένα πρωτόκολλο το οποίο σήμερα μας παρουσίασε ο συνάδελφος Ένφελτ. Η απάτη είναι κάτι που ουσιαστικά λαχιστοποιεί τα αποτελέσματα της ε, πολιτικής που έχουμε υιοθετήσει για την καταπολέμηση του καπνού και των προϊόντων καπνού. Είναι κάτι που οι νέοι, παραδείγματος χάρη, μπορεί να βρίσκουν ελκυστικό καθότι στοιχίζουν τα προϊόντα αυτά λιγότερο και την ίδια ώρα βλέπουμε τα κράτη-μέλη να χάνουν πολύ σημαντικές πηγές χρηματοδότησης. Βεβαίως και στηρίζουμε το πρωτόκολλο αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ βεβαίως και η πολιτική μου ομάδα στηρίζω αυτήν την υιοθέτηση. Την προηγούμενη εβδομάδα στην Ολομέλεια με τεράστια πλειοψηφία καταψηφίσαμε την ανανέωση της συμφωνίας ε, με την εταιρεία Philip Morris. Στείλαμε με αυτόν τον τρόπο ένα πολύ ξεκάθαρο μήνυμα προς την Επιτροπή. Πρόκειται για μια απόφαση η οποία βεβαίως ε, έχει άμεση σχέση με αυτό το πρωτόκολλο. Θέλουμε σήμερα μαζί με το Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας να δείξουμε ότι οι τυχόν συμφωνίες που συνεχίζουν να υπάρχουν με την καπνοβιομηχανία, όπως παραδείγματο χάρη αυτή που είχαμε εμείς με την Φίλιπ ε, Μόρις, σίγουρα δεν ε, μπορούν να οδηγήσουν προς μια πιο αποτελεσματική υλοποίηση της νομοθεσίας για την καταπολέμηση του καπνού και θέλουμε να πάμε προς την αντίθετη κατάσταση. Ευχαριστώ πολύ και θα δώσω το λόγο στην Επιτροπή. Δεν έχω όνομα εκπροσώπου της Επιτροπής. Ποιος θα πάρει το λόγο. Υπάρχει κάποιος από την Επιτροπή αρμόδιος για το θέμα αυτό. Είμαι από τον Όλαφ και ευχαριστώ πάρα πολύ για την στήριξή σας. Στηρίζετε την πολύ σημαντική πρωτοβουλία. Αυτό που είπε ο τελευταίος ομιλητής για την Φίλιπ Μόρις είναι πολύ σημαντικό. Ξέρουμε ότι οθετήσατε αυτήν την ε, και φυσικά νομίζω ότι η απάντηση θα σας δοθεί πολύ συγκεκριμένα για το θέμα αυτό αργότερα από την Επιτροπή. Ήσασταν πάρα πολύ σύντομος, λέει ο Πρόεδρος. Ποιος άλλος θέλει να πάρει το λόγο για το θέμα αυτό. Κανείς. Ο εισηγητής λοιπόν. Είμαι πολύ ευτυχής γιατί βλέπω ότι υπάρχει ομοφωνία όσον αφορά τη στήριξη αυτής της πρότασης. Βεβαίως δεν με εκπλήσει αυτό γιατί πρόκειται για ένα θέμα που είναι τόσο γενικό που σίγουρα διαπερνά όλες τις πολιτικές ομάδες. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ όλοι ο Πρόεδρος. 7 Απριλίου ψηφίζουμε και 20 και 21 Απριλίου θα γίνει η τελική ψηφοφορία στην Επιτροπή και τώρα περνάμε στο σημείο 10 συμφωνία με την Κολομβία και το Περού. Και βεβαίως πρόκειται για τη συζήτηση που αφορά την προσχώρηση της Κροατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θα δώσω το λόγο στον κύριο Φίσας. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Η εμπορική συμφωνία μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, και τα κράτη-μέλη και από την άλλη Κολομβίας και Περού προσυπεγράφει στις 26 Ιουνίου του 2012 και ίσχυσε μεταξύ Ευρωπαϊκής ε, Ένωσης και Περού από την 1η Μαρτίου 2013 και για την Κολομβία από την 1η Αυγούστου 2013. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 11 Σεπτεμβρίου 2012 ενέκρινε αυτή τη συμφωνία. Προβλέπεται και άλλες χώρες της κοινότητας των Άνδεων να μπορέσουν να προσχωρήσουν σε αυτή τη συμφωνία. Υπό αυτή την έννοια η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο Ισημερινός ολοκλήρωσαν τις διαπραγματεύσεις στις 11 Ιουλίου 2014 Ελπίζουμε να δοθεί τελική μορφή στη συμφωνία έτσι ώστε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να μπορέσει να εγκρίνει μέχρι τα τέλη του έτους. Απλώς θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ο δεύτερος εταίρος της κοινότητας των Άνδεων και ένας από τους βασικούς επενδυτές. Εδώ και δύο εβδομάδες είχαμε μία συνάντηση με το Monitoring Group όπου αναλύσαμε τη δεύτερη, τη δεύτερη ετήσια έκθεση για την εμπορική συμφωνία μεταξύ Κολομβίας και, με την Κολομβία και το Περού. Είναι δύσκολο να ορίσουμε ορισμένους τομείς, ε, δηλαδή οι υπηρεσίες και οι επενδυτικές ροές είναι μόνο μερικώς διαθέσιμες και η Επιτροπή θεωρεί ότι δύο χρόνια μετά τη θέση σε ισχύ συνεχίζεται η διαδικασία εφαρμογής προς ικανοποίηση όλων των μέρων. Μέσα στα πλαίσια της συμφωνίας ε, οι γενικευμένες προτιμήσεις ισχύουν. Τα απελευθερωμένα προϊόντα από το Περού και την Κολομβία έχουν αυξηθεί σημαντικά και οι, εξα... και οι εξαγωγές προς Περού και Κολομβία από Ευρωπαϊκή Ένωση. Η συμμετοχή της ε, Κροατίας είναι απόρρια της προσχώρησής της στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πρέπει η Επιτροπή και το Συμβούλιο να λάβουν τα κατάλληλα μέτρα για την συμμετοχή. Συστήνω λοιπόν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να εγκρίνει τη συμφωνία για τη συμμετοχή της Κροατίας μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, και Κροατίας και Κολομβίας και Περού. Για την περίπτωση του Ισημερινού δεν χρειάζεται ειδική συμφωνία. Θα ισχύσει αυτόματα. Έτσι έχει κατάσταση. Ευχαριστώ πολύ. Σαν Κιώδης, για τους σοσιαλιστές θα ήθελα να στηρίξω την κατεύθυνση που μας προτείνεται. Φιλελεύθερη ΙΣΙΑΡ. Α, συγγνώμη, δεν σας είδα. I have a text of um, Jan Saradil. Dear Mr. Rapporteur, dear colleagues, we agree with the rapporteur. Συμφωνούμε με τον εισηγητή. ότι η συμμετοχή της Κροατίας είναι θέμα καθαρά διαδικαστικό, νομικό το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο λοιπόν σίγουρα θα πρέπει να δώσει την έγκρισή του και να στηρίξει αυτό το επιπλέον πρωτόκολλο. Εμάς μας ε, ενησυχεί η κύρωση του πρωτόκολλου για την Κολομβία, το Περού και τον Ισημερινό, γιατί αυτό θα γίνει μόνο το Νοέμβριο ή το Δεκέμβριο του 2016 και έχω την εντύπωση ότι θα υπάρξει ένα κενό κάποιων ε, μηνών καθότι εκπνέει η συμφωνία για, την ελεύθερη, για τις ελεύθερες συναλλαγές προτιμησιακή σχέσεις με τον Ισημερινό. Θα ήθελα λοιπόν να, να μας εξηγήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τι θα συμβεί κατά τη διάρκεια αυτού του κενού αυτών των μηνών και αν υπάρχει δυνατότητα να επιταχύνουμε αυτή τη διαδικασία. Σας ευχαριστώ πολύ. Η φιλελεύθερη. Χέλμουτ. Ευχαριστώ, Μπέρντ. Εγώ συμφωνώ με τον εισηγητή, τον κύριο Φίσας. Θα ήθελα επίσης να πω ότι φυσικά η Κροατία γίνεται τμήμα αυτής της ε, συμφωνίας και σαν ένα υπεύθυνο κράτος μέλος θα πρέπει να κάνει ό,τι μπορεί έτσι ώστε να υπογραφεί το συντομότερο δυνατόν, να κυρωθεί μάλλον ε, το συντομότερο δυνατόν η συμφωνία με τον Ισημερινό ε, έτσι ώστε να μην υπάρξει αυτό το κενό. Και η Κροατία πρέπει εδώ να επιταχύνει διότι ναι, είναι ένα τεχνικό αν θέλετε θέμα, αλλά θα πρέπει να δούμε τι έχουμε πετύχει μέχρι τώρα με αυτές τις συμφωνίες, γιατί σαφώς και η κύρωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι κάτι το τεχνικό από τη μία άποψη, αλλά που έχει πολύ συγκεκριμένη πολιτική ουσία. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Έχουμε και την ακρόαση έτσι και αλλιώς για το θέμα αυτό. Σίγουρα θα πρέπει να εξετάσουμε προσεκτικά αυτό το θέμα με τον Ισημερινό. Δεν βλέπω κανέναν από τους πράσινους, ούτε από την EFTD. Ε, ο κύριος Γιώργεντσεν. Thank you very much. Ε, Ευχαριστώ πολύ. Yeah? Okay, sorry. Thank you very much. Um, well, just... Λοιπόν, σας ευχαριστώ μια μικρή παρατήρηση για την Κροατία. Να χαροποιεί το γεγονό ότι τώρα πια το ζήτημα αυτό εξετάζεται από το Κοινοβούλιο. Πράγματι είναι ένα νομικό θέμα. το οποίο πρέπει να επιληθεί. Ε, συχνά έχουμε πρόβλημα με τους ε, εταίρους μας στη Λατινική Αμερική που θεωρούν ότι σε τέτοιες διαδικασίες θα έχουν τη δυνατότητα να επαναδιαπραγματευτούν το πρωτόκολλο και Μα χαροποιεί λοιπόν το γεγονό ότι προχωράει η διαδικασία και με το Περού και σιγά σιγά θα γίνει το ίδιο και με το Μεξικό και με άλλε χώρε τη Κεντρική Αμερική. Χαίρομαι επίση που προηγήθηκε η διαδικασία με τον Ισημερινό μας ανησυχούσε ή το ενδεχόμενο να υπάρξει κενό ανάμεσα στην ημερομηνία που θα λήξει ο τρέχον κανονισμός και ε, την ημερομηνία που θα τεθεί σε εφαρμογή το πρωτόκολλο, αλλά εμείς ευελπιστούμε ότι μέχρι το τέλος της χρονιάς θα έχουν ολοκληρωθεί όλες οι διαδικασίες. Έχουμε κάνει ό,τι μπορούμε από την πλευρά μας στο επίπεδο της Επιτροπής και πολύ σύντομα θα υιοθετήσει η Κομισιόν και θα αποστείλει στο Συμβούλιο την πρότασή της για να την υπογραφεί και κύρωση του πρωτοκόλου. Μετά βέβαια η διαδικασία ξεφεύγει από το δικό μας έλεγχο, θα είναι στο, στη χέρια του Συμβουλίου, αλλά εμείς τουλάχιστον κάνουμε ό,τι μπορούμε για να φτάσει γρήγορα ε, στο Κοινοβούλιο αυτή η συμφωνία. Να, θα πρέπει να προχωρήσουμε με ταχύτητα, με ευελιξία. Αλλά βέβαια οι διαδικασίες αυτές χρειάζονται και κάποιο χρόνο. Θα προσπαθήσουμε πάντως να αποφύγουμε κενό σε αυτήν την μεταβατική περίοδο. Κύριε Βίσας. Νομίζω ότι από ευρωπαϊκής πλευράς δεν υφίσταται ζήτημα. Το είπε και ο κύριος Σόλς Απλώς θα πρέπει να διευκολύνουμε όλες τις διαδικασίες, να τις επιταχύνουμε για τον Ισημερινό, γιατί απαντώντας την ερώτηση του φοβάμαι ότι αν δεν λήξει αυτή η διαδικασία μέχρι το τέλος του έτους θα είναι δύσκολο να παρατείνουμε τη συμφωνία με τον Ισημερινό. Είναι ένα θέμα επίγον να διευκολύνουμε τις διαδικασίες. Όπως είπε και ο Χέλμουτ Σόλτς, θα μεταβούμε στον Ισημερινό. Έχουμε μια σειρά συναντήσεων και με τον Πρωθυπουργό και θα ζητήσουμε να μην γίνουν τροποποιήσεις της τελευταίας στιγμής, διότι αυτό θα πλήξει τη διαδικασία ιδιαίτερα για τον Ισημερινό. Ελπίζουμε να υπάρχει ευελιξία, ιδιαίτερα από το Συμβούλιο, και να ε, κυρώσουμε αυτή τη συμφωνία πριν από το τέλος του έτους, έτσι ώστε να μην χρειαστεί οποιαδήποτε τροποποίηση από πλευράς Κροατίας. Στην πράξη, κύριε βίζας. Έχετε δίκιο. Θα κάνουμε λοιπόν ό,τι μπορούμε. Έχουμε μια πολύ σύντομη προθεσμία για τις ε, τροπολογίες. 16 Μαρτίου στις 12, αύριο δηλαδή. Ε, τελικά όμως νομίζω δεν θα υπάρξουν και τροπολογίες, έτσι δεν είναι. Ωραία, την επόμενη συνεδρία θα ψηφίσουμε τις τροπολογίες όπως σας είπα. Και τώρα περνάμε στο σημείο 11. Λατινική Αμερική που είναι ένα τμήμα αυτής της, αυτού του πλανήτη με τον οποίο έχουμε πολύ στενές σχέσεις. Έχουμε αναφερθεί σε πολλές χώρες ήδη και η συζήτηση έχει ξεκινήσει εδώ και καιρό για την πιθανή συμφωνία μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης Μερκοσούρ είναι ένα θέμα που έχει καθυστερήσει για πολλούς ε, λόγους και προσπαθούμε να βρούμε την κατάλληλη στιγμή για να το προωθήσουμε. Ο κύριος Άλβα και εγώ έχουμε στείλει μία επιστολή, την γνωρίζετε στην Επίτροπο και θέλουμε βεβαίως να προωθήσουμε λίγο αυτή τη διαδικασία. Κύριε Σάλβα, θα σας δώσω το λόγο αμέσως. Φίξατε ορισμένα σημαντικά ζητήματα. Πρόεδρε, αποστήλαμε μία επιστολή στην Επίτροπο και προσπαθούμε να δούμε ποια οδό θα ακολουθήσουμε για να ενισχύσουμε τις ε, σχέσεις μας με το Μερκοσούρ. Υπάρχει βεβαίως η πολιτική συμφωνία καταρχήν και γι' αυτό αποτείνουμε αυτή την προφορική ερώτηση στην Επιτροπή γιατί θεωρούμε ότι το ζήτημα είναι επίκαιρο λαμβάνοντας υπόψη την οικονομική και πολιτική συγκυρία στο Μερκοσούρ. Θα πρέπει λοιπόν να ενισχύσουμε τους εμπορικούς και οικονομικούς δέσμους με αυτή τη σημαντική περιοχή του κόσμου. Η σχέση μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Μερκοσούρ είναι στρατηγικής σημασίας και για τα δύο μέρη. Γιατί και η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι σημαντική για το Μερκοσούρ και το Μπαλίν μετά από χρόνια αδιεξόδου ως προς την συμφωνία που αποτελεί νομοθετικό ορόσημο για μας θα πρέπει να προχωρήσουμε έτσι ώστε να ενισχύσουμε τους οικονομικούς και εμπορικούς δεσμούς με την περιοχή του Μερκοσούρ, αλλά και την, να δούμε και την πολιτισμική συνιστόσα. Οι οικονομικές σχέσεις έχουν μεγάλη σημασία, θα πρέπει να υποστηρίξουμε τις διαπραγματεύσεις. Η κατάσταση στο Μερκοσούρ έχει αλλάξει, η Αργεντινή έχει μια νέα κυβέρνηση και στη Βραζιλία βλέπουμε την ανησυχητική κατάσταση της κυβέρνησης. Θα πρέπει λοιπόν να επιταχύνουμε αυτές τις ε, διαγματεύσεις γιατί κάθε ανοιχτή οικονομία είναι εφημερούσα οικονομία. Αυτό ε, αφορά και την Χιλή η οποία μετά την εμπορική συμφωνία με την ε, Ευρωπαϊκή Ένωση εξάγει το διπλάσιο από ό,τι η γείτονα χώρα. Γι' αυτό θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι κάθε εμπορική συμφωνία που έχουμε επικυρώσει σημαίνει μία αύξηση των εξαγωγών της Ευρώπης προς τους εμπορικούς εταίρους. Και μην ξεχνάμε ότι αυτό σημαίνει αύξηση του ΑΕΠ και δημιουργία απασχόλησης, κάτι το οποίο απασχολεί την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό θα πρέπει να υποστηρίξουμε πολιτικά αυτές τις διαπραγματεύσεις και γι' αυτό έχει σημασία η Επιτροπή αυτή να υποστηρίξει τις διαπραγματεύσεις, διότι πρόκειται για μία ε, συμφωνία που είναι ένας πολύ σημαντικός πυλώνας για μια ενδεχόμενη ε, συμφωνία. Γι' αυτό έχουμε υποβάλει αυτή την προφορική ερώτηση. Θα θέλαμε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μας πει ποια είναι η άποψή της σε σχέση με την ε, διαπραγματεύσεων. Επίσης, ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα σε ποιους ε, τομείς μπορούμε να επιτύχουμε συνέργειες και καλύτερο συμβιβασμό καθώς και κάλυψη των καινοτόμων στοιχείων. Θα θέλαμε επίσης να ξέρουμε πώς προχωρήσαμε στα σημεία που το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κρίνει ότι θα πρέπει να προχωρήσει. Έχουμε να κάνουμε με μια στιγμή ιστορικής σημασίας που δεν μπορούμε να χάσουμε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους για την υποστήριξή σας και ιδιαίτερα τον Πρόεδρο Λάγκε και τους Σκιώδης για την συνεργασία σας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Σάλβα, θα δώσω το λόγο τώρα στους Σκιώδης, αρμόδιους για Ευχαριστώ για την παρέμβαση και για την ε, πλαισίωση αυτής της ε, προφορικής ερώτησης. Πρόκειται για ένα πολιτικό παράθυρο που ανοίγει αναπάντεχα για ε, λόγους και με παράγοντες που ορίζονται από πολλές ε, χώρες της Λατινικής Αμερικής, ιδιαίτερα μετά την αλλαγή της κυβέρνησης στην Αργεντινή. Αυτό που έχει σημασία είναι να επιτύχουμε μια εμπορική συμφωνία. Πρόκειται για έναν πολύ σημαντικό εταίρο, ποσοτικά και ποιοτικά. Βεβαίως τα τελευταία χρόνια από το 2007 και μετά έχουμε συνεχή μείωση των εμπορικών σχέσεων μεταξύ Νότιος, Νότιας Αμερικής και Ευρώπης τον ε, στην περιοχή του Μερκοσούρ. Και από πλευράς Νότιας Αμερικής υπάρχουν άλλοι εταίροι που ξεκίνησαν τέτοιες διαδικασίες. Ιδιαίτερα μετά την υπογραφή του TTIP όπου ε, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και τις διμερείς σχέσεις Κίνας-Χιλής και Κίνας-Περού. Γι' αυτό θα πρέπει να προσπαθήσουμε να φτάσουμε σε μία συμφωνία σε αυτό το χώρο όπου οι δύο μεγαλύτερες χώρες, ε, η Βραζιλία και η Αργεντινή, εκπροσωπούν και ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού. Θα πρέπει λοιπόν να λάβουμε υπόψη, όπως αναφέρθηκε σε μια συνάντηση με τον πρέσβη της Βραζιλίας, η πρόταση του Μερκοσούρ είναι μια πρόταση που έχουμε στη διάθεσή μας, αποτελεί μια ε, βάση εκκίνησης ε, πολύ καλή και υπάρχουν πολλοί παράγοντες έτσι ώστε να φτάσουμε σε μία ε, εμπορική συμφωνία. Θα πρέπει λοιπόν να διασαφινιστεί το θέμα και από εμά να δούμε ποιες είναι οι προθέσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και να δοθεί και μία όθηση του Κοινοβουλίου για να προχωρήσουμε αυτές τις ε, διαπραγματεύσεις χτες η ύπατη εκπρόσωπος είπε ότι στην, κατά τον Απρίλιο θα γίνουν ανταλλαγές προτάσεων. Θα πρέπει να είμαστε, να συμμετέχουμε σε αυτή τη συζήτηση οθώντας και τις δύο πλευρές να εξεύρουν μία λύση. Αυτό αποτελεί μία ε, σοβαρή δυνατότητα ανάπτυξης και ανάκτηση των ε, δυνάμεών μας σε αυτή την Ήπειρο που κινδυνεύουμε να χάσουμε. Ευχαριστώ πολύ. Σταμάτη. Κύριε Πρόεδρε, η ECR βεβαίως και στηρίζει αυτήν την προφορική πρόταση και είμαστε πολύ μεγάλη υπέρμαχη του να προχωρήσει αυτό το ταχύτερο δυνατόν. Θέλουμε να δημιουργήσουμε αυτήν την δυναμική. Ξέρετε ότι σήμερα η κυβέρνηση της Βραζιλίας σίγουρα δεν μπορεί να αποφύγει την περαιτέρω φιλελευθεροποίηση της οικονομίας όσον αφορά την Αργεντινή με τον νέο πρόεδρο, τον Μωρίτσιο Μάκρη, σίγουρα θα επιταχυνθεί η διαδικασία για την Συμφωνία Εμπορίου με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πιστεύω λοιπόν ότι οι περισσότερες χώρες με κροσούρ, και εδώ δεν θα αναφερθώ στην Παραγουάη, θα στηρίξουν, γιατί βλέπουν ε, πολλά ωφέλη από μια τέτοια συμφωνία μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Μερκοσούρ. Γι' αυτό και θεωρώ ότι με αυτόν τον τρόπο στηρίζουμε την ανάπτυξη, μόνο, μόνο μέσα της ανάπτυξης οι οικονομίες των χωρών αυτών μπορούν να βελτιώσουν τις επιδόσεις τους και πολύ συγκεκριμένα Κοιτάξτε παραδείγματο χάρη τι γίνεται με τον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας και ποιο θα είναι το όφελος για τους καταναλωτές μας. Εμείς θεωρούμε κάτι πάρα πολύ σημαντικό και στρέφουμε εδώ προς την Επιτροπή. Πότε πρόκειται η Επιτροπή να κινητοποιήσει αυτή τη διαδικασία και δεύτερον πόσο διατεθειμένη είναι να επεξεργαστεί με αποτελεσματικότητα και με ταχύτητα αυτήν την πρόταση, κάτι που σίγουρα μπορεί να έχει πολύ σημαντικά ε, αποτελέσματα και για την ευρωπαϊκή οικονομία αλλά και για τις επενδύσεις μας πολύ συγκεκριμένα. Ευχαριστώ πολύ για την ε, Άλτε. Ποιος θα πάρει το λόγο. Κανείς. Ο Χέλμουτ. Ευχαριστώ Μπέντ και εμείς βλέπουμε σε αυτήν την προφορική ερώτηση πολύ συγκεκριμένες ευκαιρίες για να βελτιωθούν οι σχέσεις μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών και της Μερκοσούρ. Το θέμα είναι ποια θα είναι η βάση, αν θέλετε, αυτής της διαπραγμάτευσης και ποια είναι η θέση των χωρών του Μερκοσούρα αλλά και η δική μας γιατί θυμάστε ότι πριν από 10 χρόνια ξεκίνησε η πρώτη προσπάθεια ε, διαπραγμάτευσης μιας τέτοιας συνεργασίας. Θα πρέπει σήμερα να ξαναδούμε αυτήν την ε, εντολή βεβαίως γιατί μας ενδιαφέρει εξίσου να συμπεριληφθούν και όλες οι επιμέρου διμερείς ε, συμφωνίες μέχρι τώρα νομίζω ότι δεν έχουμε λάβει σοβαρά υπόψη μας όλα αυτά τα οποία έχουν γίνει τα τελευταία 20 χρόνια θα έλεγα μεταξύ ημών και των χωρών της Λατινικής Αμερικής. Και αυτό μπορεί να προκαλέσει μια επιπλέον δυσκολία. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή γνωρίζει ότι οι χώρες του Μερκοσούρ έχουν ε, μάλλον στοχεύσει περισσότερο στη συνεργασία μεταξύ νότου-νότου. Και αναρωτιέμαι πώς θα αντιμετωπίσουν σήμερα στην πράξη οι χώρες αυτές την ε, αναζωοπήρωση, την αναγέννηση αυτής της ε, συνεργασίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Χρειαζόμαστε σίγουρα μια νέα στρατηγική, χρειαζόμαστε περισσότερη σαφήνεια και Συμφωνώ με αυτό που είπε ο κύριος ε, Ντάντι. Το θέμα των παραγωγών κρέατος ε, και γαλακτοκομικών ε, προϊόντων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το θέμα του ανταγωνισμού από την παραγωγή των χωρών αυτών. Ίσως θα πρέπει να ξαναδούμε ε, πιο συγκεκριμένα τους στόχους της COP21 και όλα αυτά να τα ενσωματώσουμε στις διαπραγματεύσεις που θα έχουμε με τις χώρες του Μεκροσούρ. Με μεγάλη ανυπομονησία θέλω να ακούσω την Επιτροπή. Ευχαριστώ πολύ. Δεν βλέπω κάποιον άλλο να θέλει να πάρει το λόγο. Θα δώσω το λόγο στην Επιτροπή. Ποιος ε, θα πάρει το λόγο. Έχω και εγώ μια ερώτηση όμως πριν απαντήσετε. Εδώ και αρκετούς ε, μήνες μιλάμε για το θέμα αυτό και <clears throat> ξέρω ότι το ίδιο θέμα συζητείται έντονα και στο Συμβούλιο. Μπορείτε να μας περιγράψετε πώς έχει η κατάσταση στο Συμβούλιο, τον συσχετισμό των δυνάμεων και πόσο έχει προχωρήσει το θέμα αυτό στο Συμβούλιο. Thank you, Chairman. And, um, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω να απαντήσω χωρίς βέβαια να προκαταλάβω την απάντηση στο προφορικό ερώτημα που θα δώσει ο Επίτροπος. Διαπιστώσαμε το ενδιαφέρον της Επιτροπής σας και την υποστήριξη που επιδεικνύεται σε αυτή τη διαδικασία διαπραγμάτευσης. Αυτό είναι ξεκάθαρο από το πολύ διεξοδικό προφορικό ερώτημα που θα υποβάλλετε. Συμφωνώ λοιπόν με πολλούς από τους ομιλητές, πολλά από τα μέλη, ότι βρισκόμαστε σε μια στιγμή όπου αλλάζουν ε, οι πολιτικές των κυβερνήσεων των χωρών του Μερκοσούρ, επομένως είναι μια κρίσιμη στιγμή την οποία μπορούμε να αξιοποιήσουμε για να προχωρήσουμε. Η Επιτροπή λοιπόν θεωρεί ότι εδώ υφίσταται μια ευκαιρία για να πετύχουμε κάτι που θέλαμε ε, εδώ και πολύ καιρό να έχουμε μια υποκοδομητική ανταλλαγή προτάσεων με αυτές τις χώρες. Και αυτό προσπαθούμε. Να συμβεί αυτό στο δυνατόν πιο σύντομα ή δυνατόν για τον Απρίλιο. Στο πλαίσιο του GPs τι επίσης γίνονται συζητήσει όπω γνωρίζετε. Και ε, ε, εκεί μέσω διαδικασία του GPC θα πρέπει να λάβουμε τι απόψει και των κρατών μελών πρώτα. Um, Σήμερα οι απαντήσεις της Επιτροπής είναι πολύ λακωνικές. Μήπως θα μπορούσατε να μας πείτε λίγα περισσότερα για το τι αναμένετε να γίνει στο Συμβούλιο και στην TPC. Και επίσης αν θεωρείτε ότι θα πρέπει να αλλάξει η εντολή διαπραγμάτευσης που έχει δοθεί στην Κομισιόν. Ναι, λοιπόν, στην TPC έχουμε τη δυνατότητα, είχαμε τη δυνατότητα μάλλον να συζητήσουμε με τους προσώπους των κρατών μελών μάλιστα και στο επίπεδο των Υπουργών τον προηγούμενο Νοέμβριο. Και στην Επιτροπή Εμπορικής Πολιτικής λοιπόν και στο επίπεδο των Υπουργών διαπιστώσαμε ότι η μεγάλη πλειονότητα των κρατών μελών υποστηρίζει την προσπάθειά μας να προχωρήσουμε σε αυτές τις ευρωγματεύσεις. Είναι ευρείες αυτές τις διαπραγματεύσεις. Καλύπτουν και πολλά θέματα και αφορούν και πολλά κράτη-μέλη. Επίσης, διαπιστώσαμε ότι τα περισσότερα κράτη-μέλη συμφωνούν με την Επιτροπή ότι χρειαζόμαστε μια συμφωνία στο τέλος η οποία θα είναι και φιλόδοξη και σωστά ισορροπημένη και ευρεία. Επίσης πολλά κράτη-μέλη υπογράμμισαν τη σημασία η πρόταση που θα μας κάνει το Μερκοσούρ να είναι υψηλής ποιότητας. Αυτό επιδιώκουμε τα τελευταία χρόνια, οι συμφωνίες μας να είναι υψηλού επίπεδου και αυτό θα προσπαθήσουμε να κάνουμε και με το Μερκοσούρ. θα έλεγα ότι τώρα έχουμε πολύ καλύτερες πιθανότητες από ό,τι στο παρελθόν να επιτύχουμε το στόχο μας. Τώρα, όσον αφορά την εντολή διαπραγμάτευση, ναι, πράγματι αυτή την είχε λάβει η Επιτροπή πριν αρκετό καιρό, αλλά εάν κάνεις το εξετάσει προσεκτικά θα διαπιστώσει ότι αναφερόμαστε σε μια comprehensive relation, σε μια ε, συνολική ε, συμφωνία ε, σχέσεων με το Μερκοσούρ, η οποία δεν θα περιοριστεί στον τομέα των εμπορικών σχέσεων μόνο, αλλά και, στην, σε άλλους τομείς όπως οι δημόσιες προμήθειες, θα υπάρχει και ένας πολιτικός τομέας, πυλώνας αν θέλετε. Επομένως είναι επαρκώς ευρεία η εντολή διαπραγμάτευσης για να αντιμετωπίσουμε, να διαπραγματευτούμε όλα τα θέματα που κατά την άποψή μας είναι απαραίτητο να συζητά κανείς επιδιώκοντας βιώσιμη ανάπτυξη. Θεωρούμε λοιπόν την εντολή διαπραγμάτευση επαρκώ ε, ευέλικτη και, και, ευρεία για να μπορέσουμε να διεξάγουμε τις διαπραγματεύσεις όπως χρειάζεται και για να περάσουμε στις διαπραγματεύσει τα μηνύματα που λαμβάνουμε από τα κράτη-μέλη στο Συμβούλιο και από το Κοινοβούλιο. Για να καταλήξουμε τελικά σε μια συμφωνία όχι ε, απαρχαιωμένη, όχι παροχημένη, που να μην περιορίζεται μόνο στα ζητήματα του εμπορίου, αλλά να είναι πιο συνολική. Αντιμετωπίζοντα και άλλα θέματα, όπως για παράδειγμα τη σύνδεση του εμπορίου με την ανάπτυξη, το δικαίωμα ε, ε, τη διαδικασία υιοθέτηση κανονιστικών πλαισίων κτλ. Ευχαριστώ. Άλλη μια ερώτηση του Μιχαήλ Ευχαριστώ. Θέλω να επανέλθω όμως σε ένα σημείο. Μιλήσατε για την εντολή. Με την κυρία Μάντρο μιλήσαμε για διαφάνεια το θέμα της διαφάνειας είναι καθοριστικό. Μας είπε ότι δεσμεύεται για όλες τις μελλοντικέ συμφωνίες να ενημερώνει το συντομότερο δυνατόν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Απ' την άλλη όμως θα πρέπει να είναι ξεκάθαρο σε αυτές τις εντολές ποιος ακριβώς κάνει τι. Δηλαδή το θέμα παραδείγματο χάρη των σημείων που συμπεριλαμβάνονται σε μια συμφωνία πρέπει να φαίνονται σε αυτήν την ενημέρωση. Παραδείγματο χάρη το θέμα της βιωσιμότητας, της βιώσιμης ανάπτυξης. Και αυτό είναι ο ρόλο τη Επιτροπής. Θα πρέπει οι πολίτε τη Ευρωπαϊκή Ένωση να καταλάβουν περί τίνο πρόκειται. Για ποιο θέμα διαπραγματεύεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με τους εταίρους μας. Και ξέρετε ότι τα τρία-τέσσερα χρόνια έχουμε διαπιστώσει ότι όταν μιλάμε για κυρίως πολιτικές συμφωνίες, ο κόσμος, οι πολίτες της Ευρώπης θέλουν να ξέρουν περί τίνος πρόκειται, για ποια θέματα και για ποια σημεία διαπραγματευόμαστε. Το θέμα λοιπόν της εντολής είναι σημαντικό. Κατά την άποψή μας, η εντολή διαπραγμάτευσης είναι παρκώς ευρεία και μας επιτρέπει να διαπραγματευτούμε για να καταλήξουμε σε μια συμφωνία η οποία θα ταιριάζει, θα είναι αντίστοιχη με τις συμφωνίες που επιτύχαμε με άλλες χώρες και με άλλους εταίρους. Και βεβαίω όλα αυτά δεν γίνονται ερήμην του Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου. Ε, παρουσιάζουμε την πρόοδο των διαπραγματεύσεων και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στην Επιτροπή Εμπορική Πολιτική και βεβαίω ε, τι απόψει που μα εκθέτετε, τι παρατηρήσει που μα κάνετε, τις λαμβάνουμε υπόψη μα στη συνέχεια των διαπραγματεύσεων. Η επιδίωξή μα είναι να αξιοποιήσουμε αυτή την εντολή διαπραγμάτευση, έτσι ώστε η τελική ε, πρόταση συμφωνία την οποία θα προτείνουμε στο Κοινοβούλιο να τύχει ε, υποστήριξη για να μην χρειαστεί να επανέλθουμε. Δεν νομίζω ότι θα υπάρξει τέτοιο πρόβλημα. Καλύπτει νομίζω η ε, εντολή διαπραγμάτευση όλα όσα χρειαζόμαστε για να συνεχίσουμε τις διαπραγματεύσεις με τις χώρες του Μερκοσούρ και να καταλήξουμε σε μια σύγχρονη συμφωνία εμπορικών σχέσεων. Μια συμφωνία που θα καλύπτει θέματα τα οποία πάντα προσπαθούμε να καλύψουμε, που έχουμε καλύψει και σε άλλες αντίστοιχες εμπορικές ε, συμφωνίες. Για παράδειγμα, όμως, οι επενδύσεις δεν καλύπτονται από την εντολή διαπραγμάτευσης, γιατί η εντολή διαπραγμάτευση αυτή είχε δοθεί πριν την συμφωνία της Λισαβόνα συνθήκη της Λισαβόνας, αλλά ταυτόχρονα γνωρίζουμε ότι οι χώρες του Μερκοσούρ δεν ενδιαφέρονται για αυτόν τον τομέα και δεν υπάρχει λόγος να περιπλέξουμε άσκοπα τις διαπραγματεύσεις. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στη διαδικασία της ανταλλαγής των προσφορών και μετά θα συζητήσουμε άμεσα με, τους, ε, με τις χώρες αυτές, με τους εταίρους μας και όταν θα έχει γίνει πρώτος γύρος ε, αυτών των ανταλλαγών και αυτών των διαπραγματεύσεων θα μπορέσουμε να έρθουμε από την πλευρά της Επιτροπής στο Κοινοβούλιο και να σας παρουσιάσουμε πιο συγκεκριμένα. Με τις επικαιροποιημένες βεβαίως ανταλλαγές προσφορών για να γνωρίζουμε ακριβώ και ποιε είναι οι θέσει του Μερκοσούρ. Παύλο, θέλετε πάλι το λόγο. Δεν έχω πολλά να προσθέσω, σύμφωνο με τον κύριο Ντάντι, γιατί ε, το Μερκοσούρ είναι ένα στρατηγικός εταίρος και αυτό θα πρέπει πάντα να το λαμβάνουμε υπόψη κατά τις ε, διαπραγματεύσεις. Ο κύριος ε, Ντάντι Μίλησε και για άλλες ε, συμφωνίες με την Αμερική, το TTIP, με τις ΗΠΑ. Αυτές οι συμφωνίες αποτελούν απόδειξη ότι πρέπει να ενισχύσουμε τους δεσμούς με αυτή την περιοχή του κόσμου και το Μερκοσούρ δεν θα πρέπει να απομονώνεται τη στιγμή που οι ΗΠΑ προωθούν διμερείς με πολλές χώρες της Λατινικής Αμερικής. Όπως είπα, το Μερκοσούρ δεν μπορεί να μείνει στην άκρη αυτής της πραγματικότητας και αυτές οι συμφωνίες θα πρέπει να ενισχυθούν με βάση μια πολιτική υποστήριξη. Ε, κύριε Ντάντι χρειάζεται μια εξισορροπημένη συμφωνία και αυτός είναι και ο στόχος μας, ο απότερος στόχος. Ο κύριος Σταβάτη ε, τόνισε αυτό που είπαμε όλοι, ότι ζούμε μία ιστορική στιγμή και αυτό δεν μπορούμε να το ξεχάσουμε. Συμφωνούμε λοιπόν για να λάβουμε υπόψη αυτό το στοιχείο. κύριος Σόλτς ε, είπε για την ανταλλαγή απόψεων με τον κύριο Γιούρκεν για την εντολή. Έχουμε εμπιστοσύνη σε αυτά που μας είπε η Επίτροπη Τέλος, ο κύριος Σόλτς μίλησε για την ανησυχία του για ορισμένα προϊόντα, ιδιαίτερα τα γαλακτοκομικά και το κρέας Ξέρω ότι πρόκειται για ευαίσθητους τομεί και θα πρέπει να λάβουμε υπόψη αυτό τον χαρακτήρα των προϊόντων κατά τις διαπραγματεύσεις. Έτσι ώστε να υπάρξει πρόοδος και να δούμε ποιες θα είναι οι επιπτώσεις αυτά τα προϊόντα που είναι σημαντικά για όλους. Σας ευχαριστώ πολύ για την υποστήριξή σας. Είναι 10, είμαστε στην ώρα μας, ακριβώς στην ώρα μας. Μπορούμε λοιπόν να περάσουμε στο σημείο 11. Πρόκειται για την ψηφοφορία Θα κάνουμε καταρχήν ε, με τις ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές μας κάρτες μια δοκιμή αρχή της ψηφοφορίας. No. No, Good. That was, that was just a test and you are in time. Κάναμε τη δοκιμή. Είμαστε και στην ώρα μας. Περνάμε στην προφορική ερώτηση για το Μερκοσούρ, σημείο 11. Αρχή της ψηφοφορίας. Πρόκειται για την κανονική ψηφοφορία αυτή τη φορά. And the vote is closed. Τέλος. Εγκρίνεται. Και τώρα θα περάσουμε στο επόμενο σημείο. Η συζήτηση για το θέμα αυτό, για την προφορική ερώτηση, θα λάβει χώρα στην Ολομέλεια. Περνάμε στο σημείο 13. Αναπτυξιακή πολιτική, συνοχή. Συμβιβαστική τροπολογία 1 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 4, τροπολογία 4 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 5 υπέρ, κατά, αποχές, Ηλεκτρονική ψηφοφορία για την τροπολογία 5. Ψηφίζουμε. Τέλος. Εγκρίνεται. 6. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 2 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 13 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 16 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 17 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 20 υπέρ κατά αποχές ηλεκτρονική για την 20 αρχή της ψηφοφορίας τέλος Η τροπολογία 20 εγκρίνεται. Συμβιβαστική 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 28 υπέρ κατά αποχές ηλεκτρονική για την 28 αρχή της ψηφοφορίας. Τέλος. Εγκρίνεται. Κατά τμήματα ψηφοφορία για την 29. Το πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Το δεύτερο. Α, όχι ελέγχουμε το πρώτο τμήμα της 29, ηλεκτρονική ψηφοφορία. Ψηφίζουμε. Τέλος. Εγκρίνεται. Το δεύτερο τμήμα της 29, υπέρ, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 30, υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται 35 σε δύο τμήματα το πρώτο υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται το δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 31 α καταπίπτει γιατί πέρασε το πρώτο τμήμα του 35. 32 υπέρ. Κατά ποχές εγκρίνεται. 33 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβιβαστική 7. Ποιος είναι υπέρ. Κατά αποχές. Εγκρίνεται. 36 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 4 ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 45 ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 49 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 5 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 53 και 54 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 55 καταπίπτει. Α, όχι ελέγχουμε ηλεκτρονικά την 53 και 54, αρχή της ψηφοφορίας. Τέλος. Εγκρίνεται. Οι υπόλοιπες καταπίπτουν. 61. Ποιος είναι υπέρ κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβιβαστική 6, ποιος είναι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 68 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 69 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται 70 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 71 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 72 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται και τώρα ψηφίζουμε για το σύνολο με ηλεκτρονική ψηφοφορία, αρχή της ψηφοφορίας. Τέλος. Εγκρίνεται. Συγχαρητήρια. Αυτό ήταν και η ψηφοφορία που είχαμε για σήμερα. Τώρα μπορούμε να περάσουμε στο σημείο 14, ε, παρακολούθηση δραστηριοτήτων των ομάδων. Έχουμε ένα επιτυχές ε, μοντέλο παρακολούθησης ομάδων και βεβαίως εδώ έχει ξεκινήσει μια διαδικασία διαπραγμάτευσης με τις διάφορες χώρες. Θα ξεκινήσω με την ομάδα παρακολούθησης για το ε, γενικευμένο σύστημα προτιμήσεων. Έχουμε ήδη συζητήσει το θέμα αυτό, όμως ε, θα δώσω το λόγο στον κύριο Φέλνερ, ο οποίος είναι και ο εισηγητής για το θέμα αυτό. I honestly uh, don't have that much. Um, to report. We've had να σας ενημερώσω για τα λίγα που έχω να σας πω. Είχαμε την συνάντηση της ομάδας εργασίας, μετά έγινε η ακρόαση, στην οποία εξετάσαμε σε μεγαλύτερο βάθος αυτά που ήδη είχαν συζητηθεί με την ε, ομάδα διοίκησης. Και αυτό ήταν όλο. is Japan. Σας ευχαριστώ. Επόμενο θέμα η Ιαπωνία. Το συζητήσαμε λίγο και χτες. Ενημερωθήκαμε για την πρόοδο. Όμως έγινε η ε, συνάντηση της ομάδας παρακολούθησης τον Ιανουάριο και θα δώσω το λόγο στον συνάδελφο να μας ενημερώσει. Πράγματι, 13 Ιανουαρίου έγινε η συνάντηση της ομάδας παρακολούθησης και εκεί ενημερωθήκαμε από τον κύριο Πετιτσάνη, ο οποίος είναι ο βασικός ε, διαπραγματευτής μας. Δεν έχει υπάρξει κάποια μεγάλη ανατροπή η ε, σημαντική εξέλιξη της διαπραγματεύσης μετά τον γύρο των διαπραγματεύσεων του Νοεμβρίου. Αυτό ήταν κάπως απογοητευτικό. Περιμένουμε ότι οι μεγάλες, τα, σημαντικά βήματα σε αυτές τις διαπραγματεύσεις θα γίνουν μετά τον, το καλοκαίρι. Η κύρωση της TTIP θα γίνει από την πλευρά της Ιαπωνίας το Ιούνιο, τέλος Ιουνίου, αρχής Ιουλίου. Και αυτό νομίζω θα διευκολύνει ε, και θα αυξήσει τις πιθανότητες μας να έχουμε θετικές εξελίξεις στο δεύτερο εξάμεινο του έτους. Τώρα, θα έχουμε περισσότερες πληροφορίε όταν ολοκληρωθεί ο 15 ο γύρος διαπραγματεύσεων. Ευχαριστώ. Και εμεί σα ευχαριστούμε από ένα θέμα Κίνα, ομάδα προβολής 28 Ιανουαρίου. Εδώ έχουμε το ζήτημα του dumping, του κατά πόσον η Κίνα ακολουθεί την οικονομία της αγοράς, Να σε ενημερώσω ότι πρόσφατα είχα και μια συνάντηση με τον ε, πρέσβη τη Κίνα. Συζητήσαμε τα θέματα χωρίς βέβαια να υπάρξει κάποια εξέλιξη. Ο κ. Μίνκλερ που είναι ο εισηγητή, δεν είναι παρόν. Μήπως κάποιο από του σκιώδεις θα ήθελε το λόγο να μας ενημερώσει. Και τώρα πάμε στι Ηνωμένε Πολιτείε δωδέκατος ο συγγνώμη, γύρος διαπραγματεύσεων με δύο ομάδες παρακολούθησης για την επεξεργασία αυτού του 12 γύρου διαπραγματεύσεων μπορεί κανείς να διαπιστώσει ότι κάτι κινείται εκεί και ότι οι θέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών σήμερα είναι λίγο πιο ευέλικτες θα έλεγα αλλά ακόμα συμφωνία δεν υπήρξε. Κυρίως συζητήθηκε το θέμα της συνεργασίας σε θέματα ρυθμιστικά, η αναγνώριση προτύπων, λίγο για τις κρατικές προμήθειες και λίγο για την προστασία των επενδύσεων, χωρίς όμως, επαναλαμβάνω, συγκεκριμένη συμφωνία. Και βεβαίως υπήρξε μία συνάντηση. Αυτήν την εβδομάδα έχουμε πάλι συνεδρίαση, όμως ε, ο χρόνος πιέζει και αν θέλουμε να πετύχουμε αποτελέσματα σίγουρα θα πρέπει να εργαστούμε πιο εντατικά και να στοχεύουμε περισσότερο συγκεκριμένα σημεία. Τώρα, το Βιετνάμ, ομάδα παρακολούθησης για το Βιετνάμ στις 16 Φεβρουαρίου θα δώσω το λόγο στον εισηγητή. Σύντομα, κύριε Πρόεδρε, ήταν η πρώτη συνάντηση μετά την υπογραφή της συμφωνίας στο τέλος του προηγούμενου έτους. Θα κάνω μια περίληψη. Ας πούμε ότι περάσαμε από ένα χρόνο επεξεργασίας ε, της ε, γλωσσικής, αν θέλετε, επεξεργασίας του κειμένου, μετάφραση, και βεβαίως ε, υπάρχει και η απόφαση που περιμένουμε από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για την συμφωνία με την Σιγκαπούρη που θα επηρεάσει τη στάση μας όσον αφορά τη συμφωνία με το Βιετνάμ. Δεν ε, προετοιμάζουμε πολλές παραπάνω συνεδριάσεις, μία στο δεύτερο εξάμεινο και βεβαίως σιγά σιγά η ομάδα αυτή θα μετατραπεί από ομάδα παρακολούθησης σε ομάδα υλοποίησης. Πρόεδρος, ευχαριστώ. Αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό, ότι περνάμε από παρακολούθηση σε εφαρμογή. Ο Καναδάς είναι το επόμενο θέμα. 23 Φεβρουαρίου ήταν η ημερομηνία συνεδρία. Σας δίνω το λόγο στον εισηγητή. Thank you, Chairman, very much. Um, ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πραγματικά. Συναντήθηκε η ομάδα προκολούθησης. Συνεχίζεται η νομική επεξεργασία των θεμάτων στο επίπεδο της Επιτροπής. Εμείς πιο συγκεκριμένα προσπαθήσαμε να συζητήσουμε συζητήσουμε ε, με τους εκπροσώπους του, του, του, το, του γεωργικού τομέα των αγροτικών προϊόντων καλωσορίζουν την συμφωνία γιατί που γνωρίζετε αυτή τη στιγμή ο αγροτικός τομέας ε, ο ευρωπαϊκός έχει πολλά προβλήματα με την εξαγωγή προϊόντων προς τον Καναδά ε, όχι μόνο που σχετικά με την τυποποίηση αλλά και άλλα. Θεωρούν λοιπόν ότι με την επίλυση των νομικών ζητημάτων θα διευκολυνθεί η δυνατότητα τους να διεισδύσουν στην καναδική αγορά. Και δεν υπάρχει πλέον καμία αμφιβολία ότι εάν δεν καταλήξει αυτή η διαπραγμάτευση στη συμφωνία μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Καναδά θα ήταν ε, αρνητικό αυτό για την ευρωπαϊκή οικονομία. Επομένως, οι ενδιαφερόμενοι αντιμετωπίζουν την προσπάθειά μας θετικά. Ευχαριστώ. 23 Φεβρουαρίου λοιπόν ήταν ε, η συνεδρίαση για τον Ισημερινό. Θα δώσω το λόγο στον κύριο Σόλτς που είναι ο εισηγητής και μετά θα μιλήσουμε και την Κολομβία. Και εγώ θα είμαι σύντομος γιατί σήμερα το απόγευμα θα συζητήσουμε το ζήτημα με τις χώρες αυτές, τις εμπορικές μας σχέσεις ε, δηλαδή και την ε, προσχώρηση του Ισημερινού στην ε, Συμφωνία ελευθέρων συναλλαγών όπως ισχύει με την Κολομβία και το Περού. Θα δούμε την προσχώρηση, το χρονοδιάγραμμα καθώς και τη δεύτερη έκθεση εφαρμογή στις συμφωνίες μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Κολομβίας ε, και Περού. Γιατί αυτό που έχει σημασία είναι να δούμε η Επιτροπή Παρακολούθησης πώς βρίσκει την φάση εφαρμογής και όπως ξέρετε απεστάλλει η συμφωνία μία εβδομάδα πριν από τις συμφωνίες του κ. Φίσας να θέλει κάτι να προσθέσει για το ζήτημα του, του, του Ισημερινού. Εμείς θεωρήσαμε ότι η διαδικασία επιτάχυνσης δεν θα πρέπει να γίνει εις βάρος της παρακολούθησης από το Κοινοβούλιο, γιατί έχουμε τις ε, προτάσεις της Επιτροπής του Συμβουλίου καθυστερούν λιγάκι και εμείς μετά πρέπει να επιταχύνουμε. Εμείς όμως θα πρέπει να έχουμε τη δυνατότητα εξέτασης αλλά φυσικά θέλουμε να επιταχύνουμε τη διαδικασία γιατί δεν θα πρέπει να ε, επιβραδύνουμε τη διαδικασία ως προς τον Ισημερινό. Ίσως ο κύριος Φίσας κάτι θέλει να πει. Ο κύριος Φίσας έχει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Όπως είπε και ο Χέλμουτ Σόλτς, είχαμε κοινή συνεδρίαση για τον ή σημερινό Περού και Κολομβία. Επειδή είναι αλληλένδετα τα ζητήματα, κρίναμε σκόπιμο να τα αντιμετωπίσουμε έτσι. Η Επιτροπή μας είπε ότι είναι δύσκολο να φτάσουμε σε συμπεράσματα, το σχολίασε προγενέστερα, γιατί με βάση τις ροές επενδύσεων δεν έχουμε στοιχεία, πλήρη στοιχεία. Η Επιτροπή όμως κρίνει ότι δύο χρόνια μετά τη θέση σε εφαρμογή η σωστή εφαρμογή συνεχίζεται προς ικανοποίηση όλων των μερών. Βεβαίως η πτώση των τιμών των αγαθών και των εμπορευμάτων οδήγησαν σε μία επιβράδυνση των ανταλλαγών. Και οι εισαγωγές και οι εξαγωγές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Περού δείχνουν μία μείωση αξιών σε σχέση με την κατάσταση στο Περού από πλευράς Κολομβίας από το 2012 μέχρι το 2014 έχουν επιταχυνθεί οι εξαγωγές, εισαγωγές. Θα ήθελα επίσης να πω ότι στην ε, Κολομβία τα εινοπνευματόδη ε, γνωρίζουν υψηλότερους ε, δασμούς σε σχέση με, τις, με τα τοπικά μπραντς. Επίσης, οι περιφερειακές αρχές της Κολομβίας επιβάλλουν περιορισμού στις εισαγωγές εινοπνευματοδών. Αυτά τα μέτρα όμως δημιουργούν ένα επιπρόσθετο κόστος για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις για τα αλκοολούχα ποτά. Άρα μειώνεται η ανταγωνιστικότητά μας στην κολομβιανή αγορά. Ε, μετά τις 13 Ιανουαρίου προσπαθήσαμε να επιλύσουμε τις διαφορές μας μέσα στα πλαίσια του ΠΟΕ. Τέλος, όταν το Κοινοβούλιο ενέκρινε την εμπορική συμφωνία με την Κολομβία και το Περού, υπήρχε πολύ σκεπτικισμός για τις πραγματικές δυνατότητες ορισμένων χωρών να αναθεωρήσουν την πορεία, του, να προβούν, τους, να προβούν σε μεταρρυθμίσεις και θεωρήσαμε ότι αυτές οι χώρες μπορούν να προωθήσουν την οικονομική ανάπτυξη με νέα μέτρα. Απόψε το απόγευμα θα μιλήσουμε γι' αυτό συμφωνώ με τον συνάδελφο Σόλτς ότι δεν θα πρέπει να απαρνηθούμε τα δικαιώματα του Κοινοβουλίου στη συμφωνία με το Εκουαδόρ. Θα πρέπει, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι αυτό θα ήταν υπερβολικό για δεύτερη φορά. Θα πρέπει να τηρήσει λοιπόν τις προθεσμίες στο Εκουαδόρ. Να προχωρήσουμε δηλαδή πολύ γρήγορα για να μην υπάρξουν προσκόμματα. Μετά έχουμε την Κεντρική Ασία. Πρόκειται ε, για τις συνθήκες ε, Εργασία στο Ουσμπεκιστάν. Ο κύριος Μορέλη δεν είναι παρόν γιατί παρακολουθεί την κατάσταση και τις εξελίξεις. Νομίζω ότι δεν είναι παρόν. Ε, γνωρίσαμε μεγάλη επιτυχία γιατί στη βαμβακοσυλλογή χρησιμοποιήθηκαν ανήλικοι. Πράγματι, κύριε Πρόεδρε, πιστεύω ότι μπορούμε να πούμε ότι την πίεση την οποία άσκησε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προς το Ουσβεκιστάν, κυρίως όσον αφορά στην εργασία των παιδιών, είχε αποτέλεσμα, μπορούμε να το διαπιστώσουμε στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εργασίας, ότι τελικά ε, έχει εξαλειφθεί η παιδική εργασία στο, στην συλλογή του Μπαμπακιού. Αλλά συνεχίζει το πρόβλημα με την εξαναγκαστική εργασία. Γνωρίζετε ότι είχαμε θίξει και τα δύο αυτά θέματα. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εργασίας έχει σε συνεργασία με την ε, σημερινή κυβέρνηση του Ουσβεκιστάν διεξαγάγει ε, έρευνες και έχουμε τις σχετικές εκθέσεις. Η κυβέρνηση έχει συνεργαστεί με τα συνδικάτα και έχουν καταλήξει σε ένα σχέδιο δράσης για την καταπολέμηση της ε, εξαναγκαστικής εργασίας. Θα πρέπει να δούμε τι θα γίνει, πώς τελικά θα εφαρμοστεί αυτό το σχέδιο δράσης κατά τη διάρκεια της περίοδου του Αυγούστου, της συλλογής του, της οδιαστό, τον Αυγούστο. Επίσης, ε, θα πρέπει να δούμε πώς το Ουσβεκιστάν θα αποδεχθεί το πρωτόκολλο για τους εργαζόμενους στον τομέα τη κλειστοφαντουργία. Αναμένουμε λοιπόν να δούμε τι θα γίνει τον Αύγουστο και έτσι έχουν τα πράγματα όσον αφορά το Ουσβεκιστάν. Λοιπόν, διαπιστώνουμε ότι ε, οι προσπάθειες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όταν είναι ε, συστηματικές, διαρκείς, έχουν αποτέλεσμα. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους λοιπόν που εργάστηκαν στο πλαίσιο των ομάδων παρακολούθησης. Και πάμε στο σημείο 15. Ε, εδώ η αρμόδια επιτροπή είναι η ΙΜΚΟ για την προστασία του καταναλωτή και το ζήτημα αναγνωματότητα σχετικά με το νομικό πλαίσιο τη Ένωση για τι τελωνιακέ παραβάσει και κυρώσει. Η δικιά μα επιτροπή βέβαια θα ασχοληθεί με την εξωτερική διάσταση του θέματο. Είναι η πρώτη φορά που συζητάει η Επιτροπή μας ε, ε, μια νομοθετική πρωτοβουλία στον τομέα αυτό. Σύμφωνα με τον κανονισμό, η Επιτροπή μας έχει αρμοδιότητα για την εξωτερική διάσταση των τελών. Είναι λογικό από τη στιγμή που ασχολούμαστε με τις συμφωνίες εμπορικών συναλλαγών. Πάντα τίθεται το ζήτημα των δασμών και των τελών. και αμέσως μετά τους δασμούς πηγαίνει κανείς και στο ζήτημα των ποινών και των προστήμων που επιβάλλονται σε περίπτωση τελωνιακής παράβασης. Επομένως λοιπόν εδώ θα πρέπει να συνεργαστούμε με την Επιτουσιακή Αρμόδια Επιτροπή, την ΙΜΚΟ και ελπίζω αυτή η συνεργασία να είναι ειλικρινής, να μην προσπαθήσει μια Επιτροπή να ε, εισβάλλει στις αρμοδιότητες της άλλης και θα δώσω τον λόγο στον εισηγητή μας για το θέμα αυτό. Αγαπητοί συνάδελφοι, πριν ακούσω το σύνολο των σχολείων σας, θα ήθελα να συναψίσω εντάχει το διάβημά μου. Όπως είπατε, η βασική μας αρμοδιότητα ως Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου είναι να δούμε την προστιθέμενη αξία της στήρισης των συμφωνιών, των διεθνών συμφωνιών. Θα πρέπει λοιπόν να το δούμε σε επίπεδο ΠΟΕ έτσι ώστε να υπάρχει συνεργασία της Τελωνιακής Ένωσης και ε, της με τους εταίρους. Αυτό σημαίνει διευκόλυνση των συναλλογών Γι' αυτό και θα δώσουμε τελική μορφή στην πρόταση της Επιτροπής έτσι ώστε να υπάρχει μία συνδεσιμότητα. Θα δείτε ότι με τις τροπολογίες 1, 5, 6 και 8 ακριβώς θέλω αυτό να κάνω, να υπάρχει μία ψαλίδα κυρώσεων γιατί αν δούμε την κατάσταση σήμερα, πώς μπορούμε να δεχτούμε να υπάρχει μια σχετική ατιμορρησία σε ορισμένες χώρες, γιατί τα στοιχεία μπορούν να αμφισβητηθούν, τα στοιχεία που προβάλλονται. Για μένα ε, δεν πρόκειται για κάτι το αναλύωτο, απλώς θα θέλουμε να δώσουμε κατευθυντήριες γραμμές στην ΙΜΚΟ, Συμβούλιο και Επιτροπή για ένα ελάχιστο και μέγιστο κοινό παρονομαστή με βάση τις τοπολογίες 1 με 3. Και αυτό σε σχέση με τον εσωτερικό μας χώρο και το συζήτησα το Φεβρουάριο στην προηγούμενη μου παρέμβαση. Μιλάμε για σχέση 1 προς 188. Θα πρέπει λοιπόν η Επιτροπή να δώσει τελική μορφή στα αριθμητικά στοιχεία, αλλά θα ήθελα να υπάρχει μια λογική στην πρότασή μου. Αυτά είναι τα σχόλια μου εν είδη εισαγωγής και θα ακούσω πολύ καλοπροαίρετα τις προτάσεις και τα σχόλιά σας. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε και η Μαρία Αρένα έχει το λόγο στη συνέχεια. Ευχαριστώ κύριε Προύστ για την εργασία σας. Το θέμα της εναρμόνισης είναι πολύ σημαντικό και αυτό που έχει σημασία είναι να ταχθούμε υπέρ των ανταλλαγών. Δέχομαι την πρόταση για το ελάχιστο και μέγιστο παρονομαστή. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι οι προτεραιότητες των αρμόδιων κρατών. Θα πρέπει να υπάρχει μια σαφήνεια στο, στις ε, διατάξεις. Επίσης θα πρέπει να υπάρχουν κυρώσεις για την αξία των εμπορευμάτων και των τελωνιακών δασμών. Εάν εισαγάγουμε αυτή τη διαφορά θα υπάρχει στρέβλωση, δηλαδή αφήνουμε το θέμα στην διακριτική ευχέρεια των κρατών. Άρα με την αναρμόνιση δημιουργούμε στρέβλωση. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε ποια θα είναι η βάση υπολογισμού με βάση το κατόφλι, το χαμηλότερο και το υψηλότερο. Στο άρθρο 11.2 και 12α θα ήθελα να πούμε ότι τα κράτη τηρούν τον κανονισμό του 2012 της 25 Οκτωβρίου 2012 σε σχέση με τις γενικευμένες δασμολογικές προτιμήσεις ε, έτσι ώστε να δούμε αυτό το ζήτημα στην ίντα γιατί υπάρχουν ε, συμφωνίες ελευθέρου εμπορίου όπου υπάρχουν και γενικευμένες προτιμήσεις. Θα πρέπει να εισαχθεί λοιπόν αυτή η έννοια στο έγγραφό σας και επειδή τα εμπορεύματα υφίστανται περιορισμούς και εποπτεία για λόγους δημόσιας ε, τάξης, ασφάλειας και υγείας, δυνάμει του άρθρου 24 παράγραφος 2 του κανονισμού, θα πρέπει να υπάρχει η ίδια αιτιολόγηση. Δηλαδή ορισμένα εμπορεύματα δεν μπορούν να μπουν στα εδάφη μας και άρα θα πρέπει να την χάνουν των ίδιων κυρώσεων. Σας ευχαριστώ πολύ όμως για την εργασία σας. Η κυρία Ντεσαρνές για το Άλτε. Σας ευχαριστώ. Πρώτα απ' όλα να πω αυτό που είχα πει και στην προηγούμενη μας συνάντηση ότι βρισκόμαστε στο ίδιο μήκο κύματο με τον εισηγητή και τον υποστηρίζουμε. Βεβαίω, η επιδίωξη τη Επιτροπής μα θα είναι μια ε, βελτίωση του σεβασμού των κανόνων του διεθνού εμπορίου. Ναι, χρειάζεται μια μεγαλύτερη εναρμόνιση του τελωνιακού του κώδικα και της τελωνιακής μας πολιτικής γιατί για να είμαστε πιο αποτελεσματικοί όχι για κανέναν άλλο λόγο δεν έχουμε διαφορετικά κανένα λόγο να εναρμονίσουμε τις πολιτικές μας. Ο στόχος είναι η αποτελεσματικότητα. Στον αφορά το ελάχιστο και το, και το μέγιστο ε, για τα πρόστιμα, συμφωνώ, είμαστε προς την σωστή κατεύθυνση. Βέβαια, ίσως θα πρέπει να δούμε ε, χρονικά πώς αυτό θα εξελιχθεί, ίσως να ξεκινήσουμε με μια γκάμα με μια ψαλίδα πιο μεγάλη η οποία σιγά σιγά να συγκλίνει. Γνωρίζουμε επίσης ότι η νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι πολύ υψηλού επίπεδου απαιτητική και στον τομέα του περιβάλλοντος και στον τομέα των εργασιακών δικαιωμάτων κτλ. Επομένως δεν θα μπορέσουμε να, να ε, υποστηρίξουμε, να, να βεβαιωθούμε ότι θα γίνεται σεβαστή αυτή η νομοθεσία αν δεν λειτουργεί εξίσου αποτελεσματικά και η τελωνιακή μας νομοθεσία. I read the text of uh, Mr. Θα διαβάσω ένα κείμενο του συναδελφού μου, ο οποίος ε, ευχαριστεί τον εισηγητή για την έκθεσή του Πρέπει να είναι προσεκτική η Ευρωπαϊκή Ένωση εξετάζοντας την θέση που θα λάβει σε αυτό το θέμα γιατί υπάρχουν διάφορα προβλήματα με την πρόταση της Επιτροπής. Πρώτα απ' όλα, όπως αναφέρει και ο εισηγητής, έγινε μια αξιολόγηση για 24 ε, πολιτικής της τελωνιακής 24 κρατών μελών, γιατί αυτή έγινε σε θελοντική βάση. Δεν μπορούμε να, να πάρουμε όμως τα, αποτελέσματα αυτής της αξιολόγησης και να τα εφαρμόσουμε και στα 28 κρατημέλη, κατά την άποψή μου. Θα ήθελα μια... την άποψη της Επιτροπής για το θέμα αυτό. Δεύτερον, υπάρχει ο κίνδυνος η Ευρωπαϊκή Ένωση να παραβιάσει τις υποχρεώσεις που έχει αναλάβει στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου με την πρόταση της Επιτροπής. Λέγεται, λέει μάλλον η πρόταση της Επιτροπής. Θα ήθελα να μου πει ο εισηγητής ποιες είναι αυτές οι συγκεκριμένε υποχρεώσεις, κάποια παραδείγματα και πώς μπορεί αυτό να διορθωθεί. Ποιε θα ήταν λοιπόν οι υποχρεώσει που έχει αναλάβει η Ευρωπαϊκή Ένωση στο ε, πλαίσιο του διεθνού δικαίου που θα μπορούσαν να τεθούν σε κίνδυνο από αυτή την πρόταση και να επισημάνουμε ότι αυτό ήταν ένα θέμα το οποίο το είχε θίξει η πολιτική μας ομάδα και την τελευταία φορά που είχε συζητηθεί αυτή η νομοθετική πρωτοβουλία, αλλά η Επιτροπή δεν μας έδωσε μια πιστική απάντηση. Αναφέρεται στο Forum Shopping. Λέγοντας ότι αυτό είναι ένας τρόπος να παρακάμψει κανείς την τελωνιακή νομοθεσία. Θα θέλαμε περισσότερες διευκρινήσεις από την πλευρά της Επιτροπής. Ευχαριστώ κύριε Προύστ για την εξαιρετική εργασία. Εμείς είμαστε κατά αυτής της πρότασης και θέλουμε να την αποσύρει η Επιτροπή. Εδώ ο τελωνιακός κώδικας επιτρέπει μια εναρμόνιση αλλά πρόκειται σαφέστατα για την ε, νομοθεσία αυτή και σε κάθε περίπτωση βασιζόμαστε σε 28 διαφορετικά νομικά συστήματα, διαφορετικές διοικητικές και νομικές παραδόσεις. Η σοβαρότητα των κυρώσεων τελικά θα διαφέρει από τη μία χώρα στην άλλη και βεβαίως εδώ θα πρέπει σαφώς βάσει της αρχής της αναλογικότητας να απορρίψουμε αυτή την πρόταση. Δεν είναι δυνατόν να εναρμονιστούν οι κυρώσεις. Και ουσιαστικά πρόκειται εδώ για αρμοδιότητες οι οποίες αρχικά ήταν ε, διαχωρισμένες, πρόκειται για αν θέλετε το ποινικό κομμάτι, το διοικητικό κομμάτι, δεν μπορούμε να τα ανακατέψουμε όλα. Και αν δεν δεχτεί να το, απορρίψει, να το αποσύρει συγγνώμη, η Επιτροπή, θα πρέπει εμείς να το απορρίψουμε. Ο κύριος Μπόχατ και εγώ θέλω να ευχαριστήσω τον εισηγητή, γιατί με ένα πολύ συγκεκριμένο τρόπο θα πρέπει να τηρηθούν οι αρμοδιότητες της ΙΝΤΑ και της ΙΜΚΟ των δύο επιτροπών. Θεωρώ ότι έχει δίκιο ο εισηγητής το ότι δεν ε, ζητάει τίποτα σε σχέση με τις κυρώσεις. Όσον αφορά τα συγκεκριμένα σημεία, εγώ δεν είμαι σίγουρος ότι έχουμε δυνατότητα να κάνουμε κάτι. Όσον αφορά το πρώτο τμήμα των τροπολογιών, την πρώτη ομάδα τροπολογιών, Υπάρχει το θέμα των διοικητικών κυρώσεων για συγκεκριμένες και ατομικές παραβάσεις. Σε αυτή την περίπτωση μπορούμε ενδεχομένως να φτάσουμε σε μία συγκεκριμένη αναρμόνιση για αυτές τις διοικητικές κυρώσεις. Όμως για το κατώτατο και το ανώτατο όριο, αν θέλετε, θα πρέπει να αποφανθεί η Επιτροπή ΙΜΚΟ, γιατί έχει πολύ περισσότερη γνώση και αρμοδιότητες για το θέμα αυτό. Τώρα, όσον αφορά την ομάδα, τη δεύτερη ομάδα τροπολογιών, συμφωνώ με την προηγούμενη ομιλήτρια. Ουσιαστικά, εδώ πρόκειται για κάτι που είναι θέμα του ΠΟΕ. Και σε αυτήν τη δεύτερη ομάδα, ομάδα τροπολογιών θεωρούμε ότι υποχρέωση έχουμε να δημιουργήσουμε μία ομοιογενή ενιαία αγορά. Και σε αυτή την περίπτωση έχουμε ξανασυζητήσει στα πλαίσια του ΠΟΕ παρόμοιες περιπτώσεις και αν στο πρώτο άρθρο της οδηγίας υπάρχει μια τέτοια υποχρέωση και όταν πρόκειται για εναρμόνιση της ενιαίας αγοράς, σε κάθε περίπτωση εδώ έχουμε την δική μας ευελιξία. Στο σημείο 3, στο άρθρο 3 της ε, οδηγίας, βλέπουμε πάλι να φύγονται θέματα που αφορούν τον ΠΟΕ και αυτή, αυτός ο συσχετισμός θα νομιμοποιούσε και θα διευκόλυνε μία υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη διευκόλυνση των εμπορικών συναλλαγών. Τα τελωνία που έχουν αρμοδιότητα για θεματα αντι anti-dumping και αυτό είναι μια σοβαρή αρμοδιότητα, σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να συμπεριληφθούν σε κάποια άλλη τροπολογία. Αυτό είναι αρμοδιότητα ΙΝΤΟ και σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να το αναλάβει ε, η Επιτροπή ΙΜΚΟ. Αυτή είναι η ε, συνολικότερη παρατήρηση που θα ήθελα να κάνω. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο Πρόεδρος. Θέλει να πάρει το λόγο η Επιτροπή. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σημειώσαμε αυτές τις ε, παρατηρήσεις. Δυστυχώς, ε, περιέργως, ο συνάδελφος από την DG Tax δεν είναι εδώ σήμερα. Σημειώσαμε όμως όλα αυτά και σαφώς θα σας ταλούν γραπτές απαντήσεις. Μπορείτε να μας εξηγήσετε γιατί δεν είναι εδώ. Δυστυχώς, Πρόεδρε, δεν γνωρίζω τους καλέσαμε για να καταλάβουμε για ποιο λόγο δεν είναι εδώ. Ζητώ συγγνώμη γιατί έπρεπε να είναι εδώ. Μπορώ να βοηθήσω την Επιτροπή. Ξέρω ότι έχουν πάει στην Επιτροπή ΙΜΚΟ. Ο συνάδελφος έφυγε από εδώ για να πάει να τους ακούσει εκεί. Υποθέτω λοιπόν ότι είναι πλέον του ενός αυτοί που εργάζονται στην Επιτροπή, στη συγκεκριμένη Γενική Διεύθυνση και νομίζω ότι δεν ε, είναι αποδεκτό κάτι τέτοιο. Δηλαδή να ασχολείται η Επιτροπή με διάφορες επιτροπές, να θέλει να είναι πανταχού παρούσα και να δείξει προτίμηση στην ΙΜΚΟ. Θα έπρεπε να παρίσταται και εδώ γιατί πρόκειται για νομοθετήματα τα οποία είναι ύψης της σημασίας. Να το διαβιβάσετε, να διαβιβάσετε αυτό το σαφές μήνυμα στην ε, ε, Επιτροπή. Ο κύριος Προύστα έχει το λόγο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους πάντες για τη συνεισφορά τους. Νομίζω ότι αυτή η έκθεση δεν έχει λήξει γιατί θα πρέπει να το εγκρίνουμε μέχρι μέσα Απριλίου και φαίνεται ότι δεν θα πρέπει να ασχοληθούμε με επικάλυψη αρμοδιοτήτων. Και όπως είπε η κυρία Ντεσαρνές, μας ενδιαφέρει η συνοχή, και η εναρμόνιση. Αυτό είπε και η κυρία Αρένα. Αυτό είναι το ζητούμενο. Για να απαντήσω στον κύριο Σταραμπάτη για τις παραβιάσεις, θα ήθελα να πω ότι οι ΙΠΑ ήδη ε, έχουν προβάλει το ζήτημα ενώπιον του ΠΟΕ. Και θα σας υπενθυμίσω αυτά που είπα την προηγούμενη φορά σε σχέση με το πρόγραμμα των τελωνίων του 2013 που δείχνουν διαφορές ως προς την εφαρμογή του πλαισίου, κάτι το οποίο πλήττει την αξιοπιστία της τελωνιακής μας ένωσης έναντι των εμπορικών εταίρων. Χρειάζεται διαφάνεια και αναγνωσιμότητα έτσι ώστε να τηρήσουμε τις υποχρεώσεις και εναντί του ΠΟΕ για να υποστηρίξουμε την αγορά μας στο σύνολό της. Όπως σας είπα, οι ΙΠΑ μίλησαν για αυτή την ε, ασυμβατότητα και γι' αυτό θα θέλαμε η πρόταση οδηγίας να εγγραφεί στα πλαίσια των διευκολύνσεων των συναλλαγών έτσι ώστε να αναλύσουμε και να συντονίσουμε χωρίς να προσκρούμε στην ε, επικουρικότητα, να τονίσουμε δηλαδή τη σημασία της επικουρικότητας, αλλά οι ανταλλαγές πληροφοριών από τον έλεγχο μέχρι την εφαρμογή χρειάζονται και για την Ευρωπαϊκή Ένωση και για τις τρίτες χώρες. Θα πρέπει να απλουστεύσουμε το σύστημα των κυρώσεων και των παραβιάσεων για να υπάρχει συνοχή. Και επιμένω ότι τα κράτη-μέλη θα πρέπει να ορίσουν τις ε, κυρώσεις όχι υπό μορφή κατοφλίου, αλλά υπό μορφή εύρους ή ψαλίδας. Σας προτείνω να τονίσουμε τον χαρακτήρα της εδαφικότητας της παραβίασης έτσι ώστε να μην γίνεται forum shopping. Στην ε, περιπτωση αντι anti-dumping για να μην υπάρχει stockpiling ε, έτσι ώστε να αποφευχθεί η καταβολή δασμών. Σε αυτό το στάδιο βρισκόμαστε. Λαμβάνω υπόψη τις προτάσεις τροπολογίας. Υπάρχει μία προθεσμία στις 18 Μαρτίου και θα συνεχίσουμε την εργασία μας επικοδομητικά και αποδοτικά ελπίζω. Στις 18 Μαρτίου είναι η προθεσμία για τις τροπολογίες στις 12 και βεβαίως 20-21 Απριλίου θα συνεχίσουμε Θα συνεχίσουμε λοιπόν με το επόμενο θέμα. Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση. Πρόκειται για τις αποφάσεις που Είχαμε πάρει τη γνωμοδότηση για την Επιτροπή Απασχόλησης καθώς και για την στρατηγική μας Trade for All. Αυτό το Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση παίζει στην στρατηγική αυτή έναν καθοριστικό ρόλο. Το Φεβρουάριο έγινε η πρώτη ανταλλαγή απόψεων και θα δώσω το λόγο στην η eh, eh, Ευχαριστώ. Πρόκειται για μια γνωμοδότηση για την ε, Επιτροπή Απασχόλησης. Εκεί θέλουμε να συμπεριλάβουμε αυτά που κατά την άποψή μας είναι σημαντικά και πρέπει να συμπεριληφθούν ε, στην έκθεση αυτή. Πολύ σύντομα λοιπόν θα σας παρουσιάσω τα σημεία αυτά. Είναι σημαντικό για μας να υπάρχει αξιολόγηση αντικτύπου για όλες τις εμπορικές συμφωνίες έτσι ώστε να γνωρίζουμε ποια είναι τα πιο ευάλωτα σημεία ή πιο ευάλωτοι τομείς. Και εδώ βεβαίως έχω πολλά επιχειρήματα υπέρ της ενίσχυσης της διαδικασίας ενημέρωσης και διαβούλευσης έτσι ώστε οι εργαζόμενοι, οι εργοδότες, οι εκπρόσωποι τους να ενημερώνονται για τις κοινωνικές συνέπειες αυτών των συμφωνιών. Αυτό που λέμε επίσης αυτήν την ε, γνωμοδότηση είναι ότι σε κάθε περίπτωση αυτό το Ταμείο για την προσαρμογή στην παγκοσμιοποίηση θα πρέπει να μπορεί να είναι προσβάσιμο για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Δηλαδή πρέπει να μειωθεί ο αριθμός των εργαζομένων μιας επιχείρησης για να, έτσι ώστε να μπορεί εκείνη να προσφύγει σε αυτό το ταμείο. Το θέμα λοιπόν του dumping είναι κάτι που συνεχίζει να μας απασχολεί. Θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν σε κάθε περίπτωση όλα αυτά τα εργαλεία για την προστασία από τις συνέπειες ε, αυτών των εμπορικών σχέσεων. Αυτή είναι η πρότασή μου. Θα δώσω το λόγο στους Κιώδης. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι να ευχαριστήσω την εισηγήτρια καταρχήν για τη γνωμοδότησή της. Αναφερόμαστε σε όλες μας τις ανησυχίες για τις συνέπειες της παγκοσμιοποίησης επί των επιχειρήσεών μας, επί της ευρωπαϊκής οικονομίας. Όπως το είχαμε πει και την πρώτη φορά που ανταλλάξαμε απόψη το θέμα αυτό, θα πρέπει να μπορούμε να προβλέπουμε τις συνέπειες αυτών των εμπορικών συμφωνιών. Και Γι' αυτό και είναι πολύ σημαντικές οι μελέτες αντικτύπου. Τα κράτη, οι επιχειρήσεις θα πρέπει να συνεργάζονται κάθε φορά για να προβλέψουν αυτές τις συνέπειες. Παράγραφος 5. Βεβαίως και στηρίζουμε τον εξυγχρονισμό των μηχανισμών προστασίας. Με αυτόν τον τρόπο θα καταπολεμήσουμε την στρέβλωση του ανταγωνισμού, κάτι που μπορεί να έχει καταστροφικές συνέπειες για τις επιχειρήσεις μας. Στην παράγραφο τέσσερα θέλω να εκφράσω εκ μέρους του ΕΛΚ κάποιες ανησυχίες. Εδώ εάν μειώσουμε υπερβολικά το κατόφλι, σε αυτή την περίπτωση ο αριθμός των ε, αιτήσεων θα αυξηθεί σε τέτοιο βαθμό που δεν θα είναι δυνατόν να ανταποκριθεί το Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση. Αυτό θεωρούμε ότι είναι κάτι που δεν μπορεί να υλοποιηθεί και σε κάθε περίπτωση θα πρέπει οι μικρομεσαίες επιχείρησεις να μπορούν να, είναι, να έχουν πρόσβαση σε αυτό το ταμείο. Γι' αυτό και θέλουμε να υπάρξουν δυνατότητες απόκλησης και εξαιρέσεων από το κατώτατο όριο. Χρειάζεται λοιπόν εδώ να βρούμε και κάποια, κάποιο τρόπο να συνδέσουμε το καθεστώς οικονομίας αγοράς των τρίτων χωρών και το Ταμείο για την Παγκοσμιοποίηση. Ευχαριστώ πολύ για την ομάδα ECR. Yeah, ναι, εγώ είμαι σαφής υπέρμαχος του ελεύθερου εμπορίου και του φιλελευθερισμού και βεβαίως θεωρώ ότι σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να πάρουμε αποφάσεις γνωρίζοντας ακριβώς την κατάσταση. Αυτό θα είναι μια πολύ σημαντική πρόοδος για την Ευρώπη. Μια ευρωπαϊκή λύση σίγουρα προϋποθέτει ενημέρωση. Και σήμερα οι δομές είναι τόσο περίπλοκες. Βλέπουμε ότι κάθε χώρα έχει τις δικές της διαρθρώσεις όσον αφορά τις προσαρμογές, τα εργαλεία προσαρμογής, τα ταμεία προσαρμογής και η ομάδα μας θεωρεί ότι βεβαίως θα πρέπει εδώ να επικρατήσει ένας ανταγωνισμός υγιής. Ευχαριστώ πολύ για τους φιλελεύθερους. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Νομίζω ότι θα πρέπει οπωσδήποτε να κρατήσουμε αυτό το ταμείο. Είναι πολύ καλό που υπάρχει, αλλά θα πρέπει να το μεταρρυθμίσουμε. Έχει μεγάλη σημασία να προτρέξουμε στην παγκοσμιοποίηση και όχι μόνο να τη διαχειριστούμε. Και για να προτρέξουμε χρειάζονται μελέτες αντικτύπου. Νομίζω ότι ο εισηγητής, η εισηγήτρια κινείται στη σωστή κατεύθυνση. Έχει μεγάλη σημασία για την αξιοπιστία του Ταμείου. Θα πρέπει να μεταρρυθμιστεί για να υπηρετεί τις ΜΜΕ. Αυτό είναι ύψης της σημασίας διότι παρέχουν εργασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση και πολλές φορές τις ξεχνάμε στην Ευρωπαϊκή Εθνική Πολιτική. Θα πρέπει λοιπόν να το λάβουμε αυτό υπόψη και να το υποστήριξουμε. Τέλος, οπωσδήποτε θα πρέπει να ενισχύσουμε τα μέσα εμπορικής υποστήριξης να κινούμαστε δηλαδή από κάτω προς τα πάνω και θα πρέπει να διαθέτουμε και μια κοινή βιομηχανική στρατηγική, κοινή στρατηγική επενδύσεων και γι' αυτό θα θέλαμε η Ευρωπαϊκή Ένωση να ανταποκριθεί και σε αυτό. Ähm, Ευχαριστώ για την ΚΟΕ. Ο κύριος Κούλογλου. Ε, Καλημέρα. Ε, ευχαριστούμε ε, την ε, εισηγήτρια για αυτήν την πολύ ενδιαφέρουσα, εξαιρετική θα έλεγα πρόταση. Είμαστε, έχουμε, είναι, αποτελεί μια ευχάριστη έκπληξη αυτή η πρόταση γιατί είναι απαραίτητο να αναγνωρίζουμε ξανά και ξανά ότι η παγκοσμιοποίηση μπορεί να έχει και αρνητικό αποτέλεσμα. Και το βλέπουμε συχνά αυτό το αποτέλεσμα στο, στο θέμα της ανεργίας και πρέπει να υπάρξουν υποστήριξη στους ανθρώπους που, ή επιχειρήσεις, στους ανθρώπους που κάνουν τη δουλειά τους και στις επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν πρόβλημα. Α, επίσης, η, Υποστηρίζω την ιδέα ότι θα πρέπει να υπάρχουν εκτιμήσεις για όλες τις εμπορικές συμφωνίες ε, και ιδιαίτερα ε, εκτιμήσεις για το αποτέλεσμα όλων των εμπορικών συμφωνιών και ιδιαίτερα στους πιο ευπαθείς ε, τομείς. Επίσης, την, επέκταση του στόχου του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση έτσι ώστε να συμπεριληφθούν ε, και εργάτες οι οποίοι έχασαν τη δουλειά τους σαν αποτέλεσμα ε, το, της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης. και πρέπει επίσης να κάθε περιοχή που μπορεί να ενταχθεί στην, ε, στην πρωτοβουλία για την νεανική απασχόληση να μπορούν ε, ε, τα, τα κράτη-μέλη ε, να προσφέρουν υπηρεσίες στους ανασφάλιστους, στους, στους άνεργους νέους. Προς το παρόν αυτό πρόκειται για μια προσωρινή ρύθμιση μέχρι το τέλος του 2017 προτείνουμε να γίνει αυτή μια μόνιμη ρύθμιση. Και υπάρχουν και δύο, τρία, τρία σημεία που θα ήθελα επιπλέον ε, να προτείνω. Πρώτον, ότι το 500, ο αριθμός 500 είναι πολύ υψηλός. Ε, θα προτείνω να πάει στους 50 ε, ε, εργαζόμενους το όριο. Έτσι ώστε να μπορούν να συμπεριληφθούν και μικρές επιχειρήσεις. Δεύτερον, ε, να, να αυξηθεί ο προϋπολογισμός για αυτό το εργαλείο από τη στιγμή που η παγκόσμια οικονομική κρίση συνεχίζεται. Ε, και το τρίτο σημείο, ε, να απλοποιήσουμε τις διαδικασίες και να ε, πληροφορήσουμε καλύτερα ε, τα κράτη-μέρη ώστε να μπορούν να συμμετέχουν στην διαδικασία αυτή. Ευχαριστώ για την προσοχή σας. Κυρία Ρένα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ την ε, Αγνές για την εργασία της για αυτό το Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση. Είναι πολύ ενδιαφέροντα τα σημεία. Αν δει κανείς πώς λειτουργεί αυτό το ταμείο σήμερα, πρόκειται για ένα ταμείο που εργάζεται και επεμβαίνει εκ των υστέρων. Όταν δηλαδή υπάρξει πλήγμα, όταν ένας ολόκληρος βιομηχανικός τομέας και κλάδος χαθεί, όταν χαθούν χιλιάδες θέσεις απασχόλησης, το Ταμείο ουσιαστικά στηρίζει κάποιους από αυτούς τους εργαζομένους για να βρουν άλλη δουλειά. Και στα πλαίσια αυτού του Ταμείου υπάρχουν πολλά αιτήματα που αφορούν μια συγκεκριμένη περιοχή. Περιοχές δηλαδή οι οποίες εγκαταλείπουν, συγγνώμη, εγκαταλείπονται από την οικονομική δραστηριότητα και τις επιχειρήσεις. Είναι λοιπόν ενδιαφέρον να δει κανεί ότι αυτές οι αιτήσει ουσιαστικά στην αρχή είναι πολλές, σιγά σιγά όμως μειώνεται με εντυπωσιακό τρόπο ο αριθμός αυτών των αιτήσεων. Γιατί, διότι ουσιαστικά πάβει να υπάρχει οικονομική δραστηριότητα σε αυτή την περιοχή. Αυτό μας δείχνουν τα οικονομικά στοιχεία. Συμφωνώ λοιπόν με την εισηγήτρια ότι θα πρέπει να υπάρξει αναθεώρηση, όπως το είπε και η κυρία Σαγνές, να υπάρξει αναθεώρηση της λειτουργίας αυτού του ταμείου. Όταν υπάρχει μια μελέτη αντικτύπου, όπως αυτή που υπάρχει σήμερα στα πλαίσια των συμφωνιών ελεύθερου εμπορίου, μια λίγο πιο προσεκτική, αν θέλετε, μελέτη αντικτύπου με συγκεκριμένα αποτελέσματα σε κλάδους δραστηριότητας και σε γεωγραφικές περιοχές. Πιο στοχευμένες δηλαδή μελέτες αντικτύπου και βάσει των αποτελεσμάτων τους το Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση θα πρέπει να μπορεί να επέμβει όχι μόνο όταν έχει γίνει το κακό, αλλά εκ των προτέρων, να υπάρξει δηλαδή μετατροπή της οικονομικής δραστηριότητας σε μία που έχει περισσότερες προοπτικές και μέλλον. Συμφωνώ επίσης ότι αυτά τα 150 εκατομμύρια το χρόνο δεν αρκούν, ιδιαίτερα αν πρέπει να αντιμετωπίσει τις επιπτώσεις της παγκοσμιοποίησης. Χρειάζεται λοιπόν αύξηση των κονδυλίων. Ευχαριστώ. Η Επιτροπή, λέει ο Πρόεδρος. Honorable Chair. Αγαπητά μέλη, πρόεδρε. I, I Ζητώ συγγνώμη, έφτασα κάπως αργά γιατί δεν ήξερα πότε θα συζητηθεί αυτό το θέμα στην ημερήσια διάταξη. Ζητώ συγγνώμη. Έχοντας αναγνώσει τη γνωμοδότηση και αφού άκουσα τις συζητήσεις όσο ήμουν παρούσα. Πιστεύω ότι αυτά που απαιτούνται από πλευρά εμπορικών συμφωνιών και των επιπτώσεών τους βρίσκονται εκτός ε, αρμοδιοτήτων του Ταμείου Αντιμετώπισης της παγκοσμιοποίησης, άρα θα πρέπει να εισαχθούν σε μελλοντικές εμπορικές συμφωνίες και σε μελέτες αντικτύπου. Έτσι θα έπρεπε να προσεγγίσουμε αυτό το θέμα. Ως προς τις ΜΜΕ, το ζήτημα αυτό έχει καλυφθεί υπό το υπάρχον ταμείο, γιατί έχουμε τομεακές και περιφερειακές περιπτώσεις και μπορούμε να μειώσουμε τον αριθμό των δικαιούχων του Ταμείου τη στιγμή που υπάρχουν σοβαρές επιπτώσεις στην ε, περιφέρεια ή την οικονομία. Μην ξεχνάτε την επικουρικότητα. Ένα τέτοιο μέσο δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί αν υπάρχουν μόνο 50 απολύσεις γιατί αυτό θεωρείται διαχειρίσιμο σε περιφερειακό ή κρατικό επίπεδο. Αν όμως τα, το κράτος είναι μικρό η περιφέρεια και η αγορά ε, εργασίας, τότε θα μπορούσε κανείς να υποβάλει αίτηση στο Ταμείο Αντιμετώπισης της ε, Παγκοσμιοποίησης και τα, το 500, ο αριθμός 500 έχει μειωθεί σε, αρκιστές, σε αρκετές περιπτώσεις όσο αφορά τους νέους ανέργους. Όπως ξέρετε, λίγη η εξαίρεση στο τέλος του επόμενου έτους και οποιαδήποτε αίτηση θα υποβληθεί τώρα θα ισχύσει μέχρι το τέλος του επόμενου έτους. Ίσως αυτό θα πρέπει να το λάβετε υπόψη. Σε σχέση με τον προϋπολογισμό, ε, αρκεί μέχρι τώρα. Αν όμως διευρυνθεί η εντολή θα πρέπει να το ξαναδούμε. Νομίζω ότι απάντησα ως προς τα ζητήματα που ανέκυψαν όσο είμαι εδώ. Δεν ξέρω αν υπάρχουν και άλλα ζητήματα που εφήγησαν εν τη απούσια μου. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ τα μέλη της Επιτροπής, καθώς και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Νομίζω ότι είναι κάτι πολύ θετικό το ότι δηλώνουμε με ευκρίνεια ότι χρειάζεται εκ των προτέρων αξιολόγηση των συνεπειών της παγκομιοποίησης παγκοσμιοποίησης και ότι οφείλουμε όχι μόνο να κάνουμε μια μακροοικονομική ανάλυση αντικτύπου, αλλά και μια μικροοικονομική μελέτη αντικτύπου, έτσι ώστε να στοχεύσουμε σωστά τα προβλήματα και τις δυσκολίες πριν αυτά συμβούν και με την συμμετοχή των εκπροσώπων, των εργαζομένων και των εργοδοτών των επιχειρήσεων για να συζητηθούν και να αντιμετωπιστούν όλες αυτές οι συνέπειες που μπορεί να προκύψουν από μια τέτοια εμπορική συμφωνία. Άκουσα την ECR που μιλάει για την ε, επικουρικότητα. Εγώ διαφωνώ με αυτό. γιατί όταν σήμερα ξέρουμε τους αριθμούς αυτών που πλήττονται, ξέρετε ότι υπάρχουν και αρκετές διαμαρτυρίες από μέρους των μικρομεσαίων επιχειρήσεων ότι δεν έχουν πρόσβαση σε αυτό το ταμείο. Πιστεύω ότι η πρόσβαση από μέρους των ε, μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε αυτό το ταμείο είναι κάτι που είναι πάρα πολύ σοβαρό θέμα. Γι' αυτό και θέλω να ξαναδούμε τα κατόφλια όσον αφορά τον αριθμό των εργαζομένων. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να απαντήσουμε με σοβαρές προτάσεις στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Εγώ δεν είχα εκφράσει άποψη όσον αφορά το μέγεθος και τα ποσά αυτού του Ταμείου και φυσικά θα εξετάσω με μεγάλη προσοχή τις προτάσεις σας. Αυτό που είναι πολύ σημαντικό είναι να έχουμε μια συγκεκριμένη πρόταση πριν ολοκληρωθεί η συμφωνία, έτσι ώστε να υπάρξει πραγματικός κοινωνικός διάλογος με την παρουσία των κοινωνικών εταίρων. Σας ευχαριστώ πολύ για την συνεισφορά σας. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο Πρόεδρος. Νομίζω ότι όντως θα πρέπει να ολοκληρώσουμε εντέρως για τη γνωμοδότησή μας στην Επιτροπή Απασχόλησης. 22 Μαρτίου είναι η προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών. Στις 6 όχι στις 12, όπως είναι συνήθως, στις 6. Άλλες 4 ώρες δηλαδή έχουμε στη διάθεσή μας. Η ψηφοφορία 21 Απριλίου έχει προβλεφθεί. Εντάξει. Ωραία. Και τώρα περνάμε στο σημείο 17. Σημαντικό σημείο, όλοι ξέρετε, ότι λόγω του πολέμου στη Συρία πολλοί άνθρωποι όπως ξέρετε περίπου η μισή, ο μισός πληθυσμός της Συρίας έχει εγκαταλείψει τη χώρα και βρίσκεται σήμερα έχουν βρει καταφύγιο σε γειτονικέ χώρες. Στην Ιορδανία, 690.000 πρόσφυγες έχουν βρει καταφύγιο σήμερα στην Ιορδανία από τη Συρία. Οι άνθρωποι αυτοί χρήζουν προστασίας και όσον αφορά την ε, ενσωμάτωσή τους στην οικονομική ζωή στις 4 Φεβρουαρίου στην συνάντηση που είχε σαν θέμα το προσφυγικό συζητήθηκε το θέμα αυτό. Η οικονομική στήριξη λοιπόν αυτών των ανθρώπων και το άνοιγμα της αγοράς, της ευρωπαϊκής αγοράς για προϊόντα που προέρχονται από τα στρατόπεδα αυτά, τους καταβλισμούς αυτούς των προσφύγων. Η Επιτροπή έχει κάποιες προτάσεις, τις οποίες θα συζητήσουμε σήμερα. Χαίρομαι ιδιαίτερα γιατί ο πρέσβης του Βασιλείου της Ιορδανίας ο δόκτωρ Ιούσεφ Μπατάνε θα έρθει και έτσι θα έχουμε και την ευκαιρία να συζητήσουμε μαζί του για όλες αυτές τις δραστηριότητες. Καταρχήν θα δώσω το λόγο στην Επιτροπή για να μας παρουσιάσει τις προτάσεις της. Uh, thank you, Mr. Chairman. Uh, Ευχαριστώ. Από ό,τι φαίνεται, σήμερα από πλευρά τη Επιτροπή έχουμε λίγο πρόβλημα με την παρουσία μα. Ε, οι συναδέλφοί μου έχουν καθυστερήσει, αλλά μου στείλαν μήνυμα ότι είναι στο δρόμο. Αυτό μονάχα μπορώ να σας πω αυτή τη στιγμή. Αν μπορούμε να περιμένουμε. So, not the best day for the commission. Όντως δεν είναι καλή μέρα για την Επιτροπή αυτή. Να διακόψουμε λοιπόν για πέντε λεπτά. Μέχρι τις και είκοσι. Okay. So, um, the commissioner is there, but now our rapporteur is gone. Έφυγε ο συγητής όμως. Πώς μπορεί κάποιος να τον φωνάξει.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 Nevertheless, so now we start. Αρχίζουμε παρόλα αυτά. Όπως εξήγησα και προηγουμένως, είμαστε εν μέσω συζήτησης για την απλοποίηση των κανόνων που αφορούν την προέλευση προϊόντων. Εδώ προϊόντων από καταβλισμούς προσφύγων με σκοπό να στηρίξουμε, να βελτιώσουμε τις συνθήκες εργασίας, να δώσουμε δυνατότητες ανάπτυξης στους ανθρώπους αυτούς που έχουν φύγει, εγκαταλείψει την εμπόλεμη Συρία και ζουν στην Ιορδανία. Ο πρέσβης της Ιορδανίας είναι εδώ μαζί μας και θα δώσω το λόγο πρώτα στην Επιτροπή και κατόπιν στον πρέσβη για να μας δώσει τη δική του άποψη για το θέμα. Ξεκινάμε όμως με την Επιτροπή, η οποία θα μας εκθέσει την πρότασή της για την απλοποίηση των κανόνων. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Καλημέρα μέρα και στα μέλη της Επιτροπής σας. Σε ευτυχείς που μας δίνετε τη δυνατότητα να ενημερώσουμε την Επιτροπή σας για αυτήν την πρωτοβουλία, την οποία έχουμε αναλάβει σε συνεργασία με την κυβέρνηση του Βασίλειου της Ιορδανίας. Ποιο είναι το πλαίσιο. Νομίζω όλοι γνωρίζουμε πόσο μεγάλο αντίκτυπο έχει η κρίση στη Συρία τις γειτονικές της χώρες. Η Ορδανία είναι μία από τις χώρες που έχει ιδιαίτερος πληγή. Σχεδόν ένα εκατομμύριο πρόσφυγες ε, Σύριοι έχουν ε, φτάσει στην Ιορδανία και ταυτόχρονα το εμπόριο που παραδοσιακά είχε η Ιορδανία με τη Συρία ε, δεν λειτουργεί πια, δεν έχει πληγή ενώ παρόλα ε, έχουν υπάρξει και προβλήματα στις εξαγωγές της Ιορδανίας προς την Τουρκία εξαιτίας των, ε, της καταστροφής των υποδομών. Η Ιορδανία έχει ζητήσει πολλές φορές από τη διεθνή κοινότητα να την βοηθήσει. Έχει απευθύνει κλήσεις επίσης προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, ζητώντας μια συνολική ε, διευθέτηση του προβλήματος των προσφύγων της Συρίας. Και ένα από τα θέματα για τα οποία ε, θα ήθελα να ενημερώσω την Επιτροπή σας είναι ότι η Ορδανία έχει ζητήσει συγκεκριμένα από την Ευρωπαϊκή Ένωση να την υποστηρίξει μέσω της πολιτικής εμπορίου. Πέρα από την βοήθεια που παρέχουμε στην Ιορδανία μέσω των πιο σχετικών πολιτικών για την αντιμετώπιση των ανθρωπιστικών καταστροφών. Η Ιορδανία έχει ζητήσει λοιπόν από την Ευρωπαϊκή Ένωση να εφαρμόζονται με μεγαλύτερη ευελιξία ε, οι κανόνες ε, για τα προϊόντα με προέλευση την Ιορδανία και άλλα μέτρα. Η Ορδανία θεωρεί ότι με αυτόν τον τρόπο θα μπορούσε να προσελκύσει επενδύσεις στη χώρα που τελικά θα οδηγήσουν σε δημιουργία θέσεων εργασίας όχι μόνο για τους ε, Σύριους πρόσφυγες, αλλά επίσης και για τους Ιορδανούς. το οποίο ίσως να ανακόψει και το ροή προσφύγων από τις χώρες αυτές, από την Ιορδανία προς ε, άλλες χώρες βορειότερα και τελικά την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τον Ιανουάριο λοιπόν του 2016 αποστήλαμε ένα ενημερωτικό έγγραφο στην Επιτροπή σας. Μια τέτοια πρόταση. και συνεχίζεται μάλλον η συζήτηση και συνεργασία με ε, την κυβέρνηση της Ιορδανίας έτσι ώστε να υποβάλει η Επιτροπή μια σχετική πρόταση Μια πιο, πιο συγκεκριμένα θα προτείνουμε ε, τροποποιήσεις στους υφιστάμενους κανόνες για την προέλευση των προϊόντων που θα έχουν συγκεκριμένο χρονική διάρκεια εφαρμογή αυτών των παρεκκλήσεων και που θα συνδέονται άμεσα με την προσφυγική κρίση. Ε, θα σας δώσω ορισμένα από τα στοιχεία που θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας στο σχεδιασμό αυτών των παρεκκλήσεων που εξετάζουμε αυτή τη στιγμή. Πρώτον, όσον αφορά τη διάρκεια. η διάρκεια πρέπει να είναι αρκετά μεγάλη ώστε να δημιουργηθούν κίνητρα για επενδύσεις, ώστε τελικά οι ε, ε, εξαγωγές της Ιορδανίας να μπορέσουν να, να κάμψουν. Γι' αυτό εξετάζουμε κάτι του τύπου 10 χρόνια, μια διάρκεια του τύπου 10 ετών, με πρόβλεψη για ενδιάμεση αξιολόγηση και πιθανώς ε, αναθεώρηση. Επίσης, θα ε, επιδιώξουμε να ορίσουμε γεωγραφικές ζώνες στο εσωτερικό της Ιορδανίας, ε, στις οποίες θα προσπαθήσουμε να ενθαρρύνουμε τις επιχειρήσεις να δημιουργήσουν θέσεις ε, εργασίας για τους πρόσφυγες. Η Ιορδανική κυβέρνηση έχει προτείνει πέντε ζώνες. Συνεργαζόμαστε μαζί τους για να καταλήξουμε στην τελική επιλογή. Πιθανώς να προσθεθούν κάποιες περιοχές, πιθανώς να αλλάξουν κάποιες περιοχές. Η Ορδανία επίσης έχει αναγνωρίσει ότι χρειάζεται ε, αυτές οι πρωτοβουλίες τελικά να οδηγήσουν σε θέσεις εργασίας για τους πρόσφυγες. Θα πρέπει λοιπόν αυτοί οι κανόνες ε, να δοθούν, να, να, που θα προταθούν στους εξαγωγείς από την Ιορδανία να είναι οι ίδιοι με εκείνους που χρησιμοποιούμε στις λιγότερο αναπτυγμένες χώρες όταν εφαρμόζεται το σύστημα του τα πάντα εκτός από όπλα. Είναι κανόνες οι οποίοι έχουν αποδείξει ότι οδηγούν σε επενδύσεις και σε ε, ε, βελτίωση του εμπορίου. Βεβαίως, προετοιμάζοντας την πρότασή μας, εξετάζουμε και τις διαδικασίες που θα ακολουθούνται για την πιστοποίηση, για την παρακολούθηση, για να είμαστε σίγουροι ότι η τελική συμφωνία θα εφαρμόζεται σωστά. Συνεργαζόμαστε επίση με την κυβέρνηση της Ιορδανία για να συμφωνήσουμε ποια προϊόντα θα καλύπτονται από, τους, από τέτοιες Λαμβάνοντας υπόψη, και τι προτεραιότητε τη Ιορδανία και το ποια προϊόντα παράγει. Γιατί διαφορετικά θα είναι απλώς διακοσμητική όποια πρωτοβουλία πρέπει να είναι τα προϊόντα που θα επιλέξουμε τα πιο σημαντικά. Εκείνα που θα οδηγήσουν σε επενδύσεις, σε αύξηση των εξαγωγών και σε θέσεις εργασίας. Τώρα τον τρόπο, όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο θα υιοθετηθεί μια τέτοια πρωτοβουλία, πιστεύουμε ότι θα μπορούσαμε να, να, να, να ληφθεί μια κοινή απόφαση της Επιτροπής ε, Σύνδεσης ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης Ιορδανίας με την οποία κοινή απόφαση θα τροποποιείται το πρωτόκολλο. Προβλέπεται μια τέτοια διαδικασία, δίνεται τέτοια αρμοδιότητα στην Επιτροπή ε, Σύνδεσης και έχει χρησιμοποιηθεί και κατά το παρελθόν με άλλες μεσογειακές χώρες. όσον αφορά την νομική διαδικασία, εδώ ε, θα κάνει πρόταση η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο λαμβάνει την απόφαση, μια και πρόκειται για θέση τη Ευρωπαϊκή Ένωση εναντί διεθνού ε, οργάνου, αλλά βεβαίω θα φροντίσουμε και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να εμπλακεί στη διαδικασία. Είναι όμω σημαντικό να κινηθούμε γρήγορα. Ε, η Επιτροπή έχει ξεκινήσει και προτίθεται, επιδιώκει μάλλον να έχει καταλήξει στην πρόταση που θα προτείνει στο Συμβούλιο τέλη Απριλίου, Αρχέ Μαΐου. Έτσι ώστε να καταλήξουμε στην κοινή απόφαση πριν ε, το τέλος του καλοκαιριού, κατά διάρκεια του καλοκαιριού. Και κλείνοντας, κύριε Πρόεδρε, προσπάθησα να σας παρουσιάσω τι, προσ... τι ε, προσπαθεί να κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στη συνεργασία με τους εταίρους μας από την Ιορδανία. ευχαριστώ να απαντήσω στις ερωτήσεις σας. Ευχαριστώ. Thanks a lot Ευχαριστώ. Ο ή μάλλον πρόεδρος ε, της ε, Επιτροπής ανάπτυξη του εμπορίου είναι εδώ. Θα δώσω το λόγο στον ε, πρέσβη. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Θα ήθελα καταρχήν να ευχαριστήσω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για το συνεχές ενδιαφέρον προς την Ιορδανία τα τελευταία χρόνια και θα ήθελα να ευχαριστήσω την έγκριτη επιτροπή σας γιατί ασχολείται με το τρέχον αυτό ζήτημα και μου δίνει την δυνατότητα να λάβω το λόγο. Ο συνάδελφος από την Επιτροπή έδωσε σαφή εικόνα για το τι συμβαίνει, μίλησε και για τεχνική υφή ζητήματα. Θα ήθελα λοιπόν να συμμεριστώ μερικές σκέψεις. Η Ορδανία κυρίες και κύριοι βρίσκεται σε μια περιοχή αρχή κλειδονισμών δείχνει όμως αντοχή και φιλοδοξίες. Προσπαθούμε να συνεισφέρουμε στις σωστές υποθέσεις και διεθνή ζητήματα. Μέσω της δραστήριες ε, διπλωματικές της δράσεις και στο Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και της Ένωσης για τη Μεσόγειο ήταν δραστήριες κτίρια υπέρμαχος κρίσιμων ζητημάτων περιφερειακού χαρακτήρα, υποστηρίζοντας ψηφοφορίες και δηλώσεις. Η Ορδανία έχει εργαστεί με εγκαρτέρηση για να υπάρξει διάλογος αποδοχή και ήταν πρότυπο ε, ανεξιθρησκείας. Αυτό αντικατοπτρίζεται και σε πολλές πρωτοβουλίες όπως το μήνυμα του ΑΜΑΝ και την Εβδομάδα Αρμονίας μεταξύ των θρησκευμάτων. Παρά τις ε, περιφερειακές κρίσεις και κλειδονισμούς, η Ορδανία εμένει στην αποφασιστικότητά της ε, για μεταρρυθμίσεις. Δεν εκμεταλλευτήκαμε αυτές τις σειράξεις στην περιοχή και με βάση το νέο νόμο για τα πολιτικά κόμματα και για τις δημοτικές αρχές προσπαθούμε να επιτελέσουμε τη σωστή πρόοδο. Ως προς τις επιπτώσεις της κρίσης στη Συρία, στην Ιορδανία, Όλοι γνωρίζετε ότι ανοίξαμε τις πόρτες μας διάπλατα σε πρόσφυγες την τελευταία δεκαετία και είχαμε συνεχείς εισρωές. Έχουμε 1,3 εκατομμύρια Σύρους οι οποίοι είναι πρόσφυγες, οι περισσότεροι ε, και ζουν σε αστικό περιβάλλον, δεν ζουν πλέον σε καταβλισμούς. Αυτό σημαίνει ότι οι πόλεις υποδοχής ε, επομίζονται το κόστος, καθώς και η κυβέρνηση. Αυτό σημαίνει μεγάλο άχθος στον ε, τομέα του ύδατος. Ήταν η τέταρτη φτωχότερη χώρα στον κόσμο και τώρα είμαστε η δεύτερη φτωχότερη ως προς τους υδάτινους πόρους, γιατί γιατί έχουμε τουλάχιστον 3 εκατομμύρια πρόσφυγες και άλλων εθνικοτήτων. Η Ορδανία είναι μια φτωχή χώρα και έχουμε και ενεργειακά προβλήματα, ειδικά μετά από την έκλειψη παροχής φυσικού αερίου από την Αίγυπτο. Επίσης το εκπαιδευτικό σύστημα έχει πληγεί, δουλεύουν διπλό και τρίπλο βάρδια οι καθηγητές και οι δάσκαλοι, καθώς και το διοικητικό προσωπικό. Προσπαθούμε να συμμετέχουν τα παιδιά των σύρων στα σχολεία, αλλά τα όρια μας είναι αυτά που είναι. Υπάρχουν όρια τα οποία δεν μπορούμε να υπερβούμε. Δεν μπορούν όλα τα παιδιά να μπουν στο σχολείο. Το σύστημα υγείας έχει πληγεί επίσης γιατί όλοι οι Σύροι θα πρέπει να έχουν πρόσβαση στη δημόσια υγεία όπως και όλοι οι Ορτανοί. Αυτό σημαίνει μεγάλο φόρτο για μας, γιατί ένας Ιορτανός μπορούσε να πάει σε μια κλινική και να έχει μέση αναμονή 20 λεπτά. Τώρα έχει 3 με 4 ώρες. Επίσης και στην απασχόληση το θέμα είναι επικίνδυνο. Η Σύριοι στην Ιορδανία, η Ορδανία έχουν καταλάβει 170.000 θέσεις. Κάθε θέση εσύ για έναν πατέρα πενταμελούς οικογένειας. Αν ε, το πολλαπλασιάσετε επί 175.000 φτάνουμε στο 1 εκατομμύριο. Άρα οι, οι Ορδανοί έχουν μειωμένα εισοδήματα. Επιπρόσθετα έχουμε 400.000 Ιρακινούς μετά τον ε, πόλεμο του κόλπου δεν είναι πλέον πρόσφυγες, αλλά χρησιμοποιούν όλες τις υποδομές, ε, το, τους υδάτινους πόρους, την εκπαίδευση, την υγεία και ούτω καθεξής. Και επειδή έχουμε μεγάλη ανέξη θρησκεία, έχουμε δεκάδες χιλιάδες χριστιανούς και γεζίδι οι οποίοι υφίσταντο την πίεση και την βία της ΔΑΕΣ και έτσι επιμερίζουμε τους πολύ μικρούς και περιορισμένους πόρους μας. Τα τελευταία χρόνια είχαμε ε, γεμενίτες και ε, ε, Λίβιους, τουλάχιστον 100.000 που προσήλθαν, ακριβώς γιατί είμαστε μια ανοιχτή κοινωνία, είμαστε πολύ ανεκτικοί, αλλά όπως είπε και η, αυτή, αυτού μεγαλειώτης ο βασιλιάς, έχουμε φτάσει σε ένα σημείο βρασμού. Άρα τα τελευταία 17 ε, χρόνια προσπαθούμε να βοηθήσουμε τους πρόσφυγες. Έχουμε μία μεγάλη παράδοση, αλλά η διεθνής κοινότητα μας έδωσε μόνο το 36% από τις συνολικές ανάγκες μας τα τελευταία δύο χρόνια. και το υπόλοιπο 70% πρέπει να καλυφθεί από την κυβέρνηση της Ιορδανίας. Το κόστος επί του προϋπολογισμού ήταν 7 δις δολάρια το 2011. Το νέο σχέδιο 16-18 χρειάζεται 8 δις δολάρια Αμερικής. Η Ορδανία προσπαθεί να βοηθήσει τους εταίρους στα, στην ε, ε, Ένωση για να μην υπάρχουν υπερβολικές ροές στην Ευρώπη και καταβάλει κάθε προσπάθεια να σταματήσει τη ριζοσπαστικοποίηση και την τρομοκρατία καθώς και τους ξένους μαχητές που θέλουν να μεταβούν στην Ευρώπη. Ήμασταν πάντα αξιόπιστος εταίρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι αναταραχές στην περιφέρεια έχουν μεγάλες επιπτώσεις, όπως είπε και ο συνάδελφος της Κομισιόν. η παραδοσιακή εμπορική δρόμοι και διάβλοι έχουν χαθεί, κάτι το οποίο προσθέτει και πλήττει τους πενιχρούς πόρους που έχει ο προϋπολογισμός μας. Η Ορδανία λοιπόν αποφάσισε να προβάλλει στη διεθνή κοινότητα μία πολύ θαραλέα ολιστική προσέγγιση, διότι οι μετανάστες δεν θα επιστρέψουν στα σπίτια τους. Εμείς προσπαθήσαμε να τους κάνουμε να νιώσουν χρήσιμοι, να έχουν μία σταθερότητα, για να μην αναλάβουν αυτό το επικίνδυνο ταξίδι προς τη Δύση. Σύμφωνα με μία έρευνα της ΥΠΑ, της ε, ε, εποπτείας για τους πρόσφυγες, είπα της αρμοστίας με συγχωρείτε για τους πρόσφυγες, ε, φαίνεται ότι η Ορανδανία προσπάθησε να συνεργαστεί με τη διεθνή κοινότητα και μερικοί φίλοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση δυστυχώς μας είπαν ότι θα πρέπει να αποστείλουμε πλέον ε, πρόσφυγες προς την Ευρώπη. Τους ευχαριστήσαμε και είπαμε ότι εμείς δεν εκβιάζουμε, δεν εκμεταλλευτήκαμε ποτέ κρίσεις, γι' αυτό προσπαθούμε να συνεργαστούμε με τους εταίρους για να βρούμε λύσεις και να παραμείνουν οι Σύριοι στην Ιορδανία. Γι' αυτό δημιουργήσαμε 100 με 200 χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας ανάλογα με τις επενδύσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση και βεβαίως όλα αυτά εξαρτώνται από το πόσο μπορούμε να φτάσουμε σε μια συμφωνία με τους εταίρους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό μιλάμε για πέντε ε, βιομηχανικές ζώνες όπου να συμμετέχουν και Σύριοι μαζί με τους Ιορδανούς και θα προβάλλουμε και νέες αγορές όταν ε, φτάσουμε στο σημείο εξαγωγών. Είχαμε δυσκολίες στις διαπραγματεύσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Επιτροπή Εμπορίου σε σχέση με τους ε, κανόνες προέλευσης και τις προμήθειες γι' αυτό και προσφέραμε αυτό το σχέδιο. Ζητήσαμε μία διευκόλυνση 15 ετούς διάρκειας για τους κανόνες προέλευσης όπως ισχύει για τον Καναδά και τη ΣΥΠΑ μιλήσαμε για μία προστιθέμενη αξία κατά 35% αλλά από τη Γενική Διεύθυνση Εμπορίου μας πρόβαλαν την προσέγγιση των λιγότερο αναπτυγμένων χωρών. Είναι δεκαετής η προσφορά και θα αναθεωρηθεί μετά από πέντε χρόνια θα πρέπει να πείσουμε τους επενδυτές να προσέλθουν. Γιατί τα δέκα χρόνια, η δεκαετία δεν είναι και μια τόσο μακρά περίοδος. Νομίζω ότι θα σταματήσω εδώ και οποιαδήποτε ερώτηση είναι πρόσδεκτη. Ο κύριος Μορέλ, ο μόνιμος εισηγητής, έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τον Πρέσβη για τη μαρτυρία του και για τις παρατηρήσεις. Πρόκειται για κάτι που δεν είναι εμπορικό, πρόκειται για μια πολιτική εταιρική σχέση που καλούμαστε να συνάψουμε με μια χώρα η οποία έχει πληγεί άμεσα από την Συριακή κρίση, μια χώρα που πραγματικά υποδέχεται χιλιάδες πρόσφυγες. Αν κοιτάξει κανείς τι γίνεται στην Τινησία, στην Ιορδανία, το Λίβανο, θα πρέπει και εμείς να αναρωτηθούμε τι κάνουμε για να υποδεχτούμε πρόσφυγες. Πρόκειται για πολύ σημαντικές αναταράξεις από δημογραφικής απόψεως αλλά και οικονομικής. Η Ιορδανία παραδοσιακά έκανε εξαγωγές προς την Συριακή αγορά. Αυτό λοιπόν είναι κάτι που σαφώς θα πρέπει να οδηγεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε περισσότερη αλληλεγγύη. Και από μακροοικονομικής απόψεως και βεβαίως κάθε άλλη λύση θα πρέπει να εξεταστεί σε διμερές και πολυμερές επίπεδο. Η διεθνής κοινότητα το Φεβρουάριο δεσμεύθηκε στο Λονδίνο έτσι ώστε να υπάρξει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο υποστήριξης της Ιορδανίας και με επιμέρους μέτρα πολύ σημαντικά για μας, για την Επιτροπή μας. Η Ιορδανία έχει υποβάλει μια αίτηση για την ε, πιο ευέλικτη αντιμετώπιση των ε, εισαγωγών από την ε, Ιορδανία, ιδιαίτερα σε κάποιες συγκεκριμένες περιοχές, ε, ζώνες ειδικών επενδύσεων όπως το ονομάζουν, οι περισσότεροι πρόσφυγες, όπως μας λέει, ακούσατε τον κύριο Πρέσβη, δεν ζουν πλέον σε καταβλισμούς, αλλά σε αστικές περιοχές, σε γειτονιές, με τους υπόλοιπους πολίτες της Ιορδανίας. Αυτοί λοιπόν οι κανόνες, κανόνες προέλευσης σε ποσοστά 35% που ισχύει για τον Καναδά και τις Ηνωμένες Πολιτείες δεν μπορεί να ισχύσει στην περίπτωση ε, της Ιορδανίας. Χρειάζεται λοιπόν επέκταση, διεύρυνση με κάποιους περιορισμούς χρονικούς, βεβαίως γεωγραφικούς, θα πρέπει να επιλέξουμε προϊόντα που είναι ε, καθοριστικά για την ανάπτυξη στην Ιορδανία, είτε προϊόντα που κατασκευάζονται από πρόσφυγες. Η Ιορδανία δεν έχει υπογράψει την Σύμβαση της Γενέβης, παρόλα αυτά επιτρέπει στους πρόσφυγες να συμμετάσχουν στην ε, αγορά εργασίας της Ιορδανίας με πρότυπα που βρίσκονται στα επίπεδα του Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση λοιπόν καλείται εδώ να στηρίξει μια χώρα η οποία με τέτοια ταχύτητα και αποτελεσματικότητα ανταποκρίθηκε σε αυτό το κύμα ε, προσφύγων και εμείς θα πρέπει να δείξουμε αλληλεγγύη. Ευχαριστώ πολύ. Σκιώδη συζήτηση, η κυρία Ντεσαγνέζ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Συμφωνώ πλήρως με τον εισηγητή. Τα ίδια πιστεύουμε και εμείς. Ακούσαμε τον πρέσβη με μεγάλο ενδιαφέρον. Αντιλαμβανόμαστε πόσο μεγάλη είναι αυτή η πρόκληση, πόσο δύσκολο είναι για τη χώρα του να αντιμετωπίσει το πρόβλημα, αλλά μην ξεχνάμε ότι πρώτα απ' όλα, πρώτοι, πρώτοι αυτοί που έχουν ε, ένα τεράστιο πρόβλημα να αντιμετωπίσουν είναι οι ίδιοι οι πρόσφυγες από τη Συρία που εγκατέλειψαν τις αιστείες τους. Φυσικά είναι δύσκολο και για τις χώρες υποδοχής. Αντιλαμβάνομαι ε, κύριε Πρέσβη ότι υπάρχουν προβλήματα στη χώρα σας με, με το, το ζήτημα της του ότι οι πρόσφυγε χρειάζονται του ίδιου πόρου με τους πολίτες μιας χώρας. Και εμένα αυτό μου θυμίζει πόσο δεν έχουμε συζητήσει το θέμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πόσο ε, δίνουμε υποσχέσει ή κάνουμε σχέδια, λαμβάνουμε αποφάσει και στην πράξη δεν γίνεται τίποτα. Επομένω, πραγματικά θα έπρεπε η Ευρωπαϊκή Ένωση να ανταποκριθεί και να σταθεί στο ύψο των περιστάσεων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να βοηθήσει με όλους τους τρόπους που έχει στη διάθεση της, ε, τις που υποδέχονται τους ε, πρόσφυγες, διορθώνει τον εαυτό της όχι του μετανάστε του Σύρους πρόσφυγες και γι' αυτό το λόγο πιστεύω ότι η πρόταση της Επιτροπής είναι προς τη σωστή κατεύθυνση γιατί πρέπει να δώσουμε κάποιες προοπτικές για το μέλλον στους Σύρους πρόσφυγες που βρίσκονται στη χώρα σας. Βεβαίως πρέπει να οδηγηθούμε προς μια σταθερότητα, να, να βοηθήσουν την Ιορδανία να διατηρήσει τη σταθερότητα της μάλλον με αυτή την ε, εισρωή προσφύγων και ε, Βεβαίω, συμφωνώ και με αυτό που είπε ο εισηγητή κ. Μορέλ, ότι ναι, χρειάζεται, ε, χρειάζονται κάποιοι περιορισμοί χρονικοί όσον αφορά τα προϊόντα, αλλά να είναι τέτοιοι οι περιορισμοί που και να είναι αρκετά μακρά η διάρκεια των παρεκκλήσεων, αλλά και να αφορά και τα προϊόντα εκείνα που θα δημιουργήσουν τις θέσεις εργασίας. Γιατί πραγματικά η Ιορδανία έχει αναλάβει περισσότερα από όσο τις αναλογούσαν με αυτήν την κρίση και με αυτή τη σύγκρουση. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων, όπως είπα. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε, Λίντα. Ε, Λίντα, μάλλον, έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ. Και σας ευχαριστώ και την πρόσκληση. Κύριε Πρέσβη, πραγματικά θα ήθελα να ήταν περισσότεροι συνάδελφοι παρόντες για να ακούσουν αυτά που μας είπατε, γιατί πιστεύω ότι πολλοί, πολλά μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που δεν έχουν επισκεφτεί ούτε την Ιορδανία, ούτε την Τουρκία, ούτε την Νότια Τουρκία, δεν γνωρίζουν τι συμβαίνει. Δεν έχουν δει αυτές τις περιοχές όπου, ε, που έχουν υποδεχθεί πολλούς πρόσφυγες και όπως είπατε δεν ζουν όλοι σε καταβλισμούς. Αυτές οι χώρες λοιπόν αντιμετωπίζουν τεράστιες τεράστια προβλήματα, τεράστιες προκλήσεις στην προσπάθειά τους να ενσωματώσουν, να υποδεχτούν τους πρόσφυγες. Επομένω, α μην ξεχνάμε ότι οι περισσότεροι πρόσφυγε από αυτή τη σύγκρουση στη Συρία βρίσκονται όχι στι πλούσιε χώρε, αλλά στι αναπτυσσόμενες χώρε σε χώρε μέσου εισοδήματο όπω η Ορδανία. Και όπω και οι συνάδελφοί μου, αισθάνομαι ότι πρέπει να προσεγγίσω το θέμα με μια κάποια ταπεινότητα, βλέποντα τι κάνει μια χώρα όπω η Ορδανία σε σχέση με αυτά που θα έπρεπε να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να αξιοποιήσει ε, όλα τα εργαλεία που έχει στη διάθεσή τη, είτε είναι ο προπολογισμό για την αναπτυξιακή βοήθεια ή άλλα εργαλεία, για να βοηθήσει όλε αυτέ τι χώρε. Γιατί η κρίση διαρκεί και μπορούμε εύλογα να αναμένουμε ότι οι πρόσφυγες εγκαταλείπουν τη χώρα τους και θα παραμείνουν για πολλά χρόνια εκτός της χώρας τους, είχα γνωρίσει πρόσφατα έναν πρόσφυγα από την Σομαλία, ο οποίο έχασε όλη του την πρωτοβάθμια εκπαίδευση, τη δυνατότητα να έχει πρωτοβάθμια εκπαίδευση, γιατί έφυγε από την αιστεία του όταν ήταν 9 χρονών και έζησε 14 χρόνια σε καταβλισμό. Άρα, χρειάζεται να αλλάξουμε τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα αυτό. Χρειάζεται να έχουμε μια προσέγγιση πιο μακροπρόθεσμη θα ήθελα να ακούσω την πλευρά της Επιτροπής, τι σκοπεύει να κάνει και η ΕΚΟ. Καλωσορίζω την συμφωνία με την Ιορδανία που συνήθισε στο Λονδίνο. Αναρωτιέμαι, μόνο μπορώ να φανταστώ πόσο ε, δύσκολο θα είναι όταν ξεκινήσει ε, η Ορδανία να δίνει άδειε εργασίε στου πρόσφυγε από τη Συρία, όταν σκέφτομαι τι συμβαίνει στη χώρα μου, όταν συζητάμε για το δικαίωμα στην εργασία των προσφύγων. Ε, Επομένω, πρέπει να του υποστηρίξουμε όσο μπορούμε. Κύριε Πρέσβη, θα ήθελα να σα ρωτήσω για τα εξή. υπάρχουν πρόσφυγες εγκλωβισμένοι στα σύνορα θα ήθελα περισσότερες ε, πληροφορίες για αυτό. Βέβαια έχουμε παρόμοιες καταστάσεις στην Ελλάδα. Ε, πριν λίγο ήμουν σε μια συνάντηση και άκουσα για τους ε, πρόσφυγες που βρίσκονται εγκλωβισμένες στα, σύνορα με, στα βόρεια σύνορα της Ελλάδας. Το ζήτημα λοιπόν αυτό πρέπει να αντιμετωπίσουμε όχι μόνο στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά συνεργασία και με τους εταίρους μας για να βοηθήσουμε ο ένας τον άλλον να ξεπεράσουμε αυτή τη δύσκολη κρίση. Ελπίζω λοιπόν να συμφωνήσουμε και να βρούμε μακροπρόθεσμες λύσεις. Ευχαριστούμε. Thanks, I'll be brief, but I to speak. Θα είμαι σύντομο, αλλά παρά το γεγονός δεν έχω να, προσθέσει, να προσθέσω πληροφορίες. Από το 2013, από τις εκλογές στην Ιορδανία, ήμουν παρατηρητής. Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη λοιπόν ότι το 2013 κάτω από κατά δύσκολες ε, καταστάσεις, η Ορδανία διενέργησε ελεύθερες και ειρηνικές εκλογές. Βεβαίως ε, μιλήσαμε για τη βελτίωση του συστήματος τότε, όμως είναι μια σταθερή δημοκρατία σε μια περιοχή που δεν φημίζεται για κάτι τέτοιο. Αυτό θα πρέπει να διατηρηθεί και να εκτιμηθεί. Βεβαίως ξέρω ότι έχει αυξηθεί δραματικά ο αριθμός των προσφύγων, αλλά ήδη το 2013 υπήρχαν πολλοί πρόσφυγες ε, στην Ιορδανία. Επισκέφθηκα διάφορα μέρη της Ιορδανίας τέσσερις με έξι φορές και μου έκανε μεγάλη εντύπωση η, ε, ε η, το μέτρο και η έλλειψη αμετροέπειας που έδειξαν οι Ιορδανοί. Και όπως είπε και η Λίντα, ίσως γι' αυτό το λόγο δεν δώσαμε σημασία στην Ιορδανία όσο θα έπρεπε, επειδή είναι ανεξίθρισκη, δεν έχει φυσικούς πόρους. Δηλαδή προσπαθεί να φτιάξει και να πουλά πράγματα. Μιλήσαμε και για τους, τις εμπορικές οδούς που έχουν καταστραφεί, όπως είπε και ο πρέσβης το 2013 είχε ζητηθεί να αλλάξουμε τους κανόνες προέλευσης και δυστυχώς τότε προσκρούσαμε σε έναν τοίχο. Έκτοτε έχουν αλλάξει τα πράγματα, δεν ξέρω πότε ακριβώς, αλλά όπως είπε και η Λίντα, στη διάσκεψη του Λονδίνου ε, δόθηκε, δόθηκε μία όθηση ο Καναδάς και η ΙΠΑ έχουν ένα 60% συσσόρευση κανόνων προέλευσης. Εμείς μπορούμε να επιταχύνουμε την αλλαγή αυτή γιατί είναι επίγουσα. Αυτό θα ήταν μια σημαντική ε, συνεισφορά Εάν λάβουμε υπόψη την κλίμακα του προβλήματος, αυτά που έχουμε παραχωρήσει δεν αρκούν. Ευχαριστώ. Η Επιτροπή. Θα σας ξαναδώσω το λόγο. Αυτό που είπε ο Ντέιβιτ είναι πολύ σημαντικό και αφορά τη συσσόρευση τέτοιων κανόνων προέλευσης και κοιτώντας μια απλοποιημένη διαδικασία μπορεί κανείς να πει ότι εν ώψη αυτών των τόσο σημαντικών προκλήσεων ίσως θα πρέπει για να ξεπεραστούν αυτές οι προκλήσεις και αυτές οι δυσκολίες να τους παρέχουμε ε, ένα τελείως διαφορετικό καθεστώς. Τώρα, το θέμα των επενδύσεων. Σε όλες τις συμφωνίες, τις επενδυτικές, αλλά και τις εμπορικές συμφωνίες που έχουν μία πτυχή επενδύσεων, προβλέπουμε 20 χρόνια. Δηλαδή η απόσβεση αυτών των επενδύσεων ουσιαστικά προβλέπεται να έχει ολοκληρωθεί σε αυτήν την 20 Τώρα, μιλάμε για 10 χρόνια. Γιατί, μπορείτε να μας πείτε. Και να μας εξηγήσετε και λίγο πιο συγκεκριμένα ποια είναι τα προϊόντα αυτά τα οποία στοχεύει η πρότασή σας. Κάτι δηλαδή που δεν θα προκαλέσει συγκεκριμένα προβλήματα και δυσκολίες ε, στην ευρωπαϊκή οικονομία. Ευχαριστώ Πρόεδρε να ευχαριστήσω και τα μέλη της Επιτροπής για την όθηση και τη στήριξη που μας δίνουν. Άκουσα πολύ θετικά σχόλια και φυσικά θα συνεχίσουμε τις προσπάθειές μας έτσι ώστε να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε αυτήν την συμφωνία όσο συντομότερο γίνεται. Πριν το καλοκαίρι ελπίζουμε να έχουν γίνει τα πρώτα σημαντικά βήματα. Ο πρέσβης της Ιορδανίας αναφέρθηκε στις διαπραγματεύσεις για μια γενικότερη συμφωνία ελεύθερου εμπορίου. Πρόκειται για μια διαδικασία όμως που θα πάρει πολύ περισσότερο χρόνο. Συνεχίζουμε να επεξεργαζόμαστε το θέμα αυτό με την Ιορδανία Λαμβάνοντας υπόψη όλα αυτά τα σημεία που έθιξε ο πρέσβης όπως τις δημόσιες προμήθειες κτλ. Όσον αφορά τώρα τους κανόνες προέλευσης, την απλοποίηση, αλλά και το χρονοδιάγραμμα, την προθεσμία, είχαμε σκεφτεί ακόμα πιο σύντομα, ακόμα πιο μικρή χρονική περίοδο από τη δεκαετία κύριε Πρόεδρε, καταρχήν. Και αυτό το... Η δεκαετία ουσιαστικά είναι ένα είδος ε, εξισορροπημένης πρότασης μεταξύ της αρχικής και της εικοσαετίας. Κάτι που θα μπορούσε να περάσει στο Συμβούλιο. Δεν έχω συγκεκριμένες άλλες νομίζω απαντήσεις να δώσω. Θα ήθελα να σας διαβεβαιώσω, θα συνεχίσουμε την επεξεργασία του θέματος και θα ενημερώσουμε την Επιτροπή για περαιτέρω πρόοδο στο θέμα αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Πότε μπορείτε να υποβάλλετε τη συγκεκριμένη πρόταση. Η πρόθεσή μας είναι να ολοκληρώσουμε την πρότασή μας έως τις αρχές Μαΐου. Τέλος Απριλίου, αρχές Μαΐου και να υποβάλουμε ε, την πρόταση αυτή στο Συμβούλιο έτσι ώστε να υπάρξει πριν το καλοκαίρι μια κοινή απόφαση Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, Ιορδανίας. Ταυτόχρονα συνεχίζουμε τις επαφές μας με τις αρχές της Ιορδανίας. Ταυτόχρονα δηλαδή με αυτά που γίνονται εδώ στο εσωτερικό της Επιτροπής. Θέλουμε πραγματικά να ενισχύσουμε όλες αυτές τις πρόπτικες που θέλει η Ορδανία να δώσει στους πρόσφυγες. Ναι, νομίζω ότι είναι σημαντικό, λέει ο πρόεδρος, να επιταχυνθεί η διαδικασία και να πιέσουμε λίγο και στο Συμβούλιο να επιταχυνθεί η διαδικασία. Έχετε το λόγο κύριε Πρέσβη. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω όλους για τα θετικά σας σχόλια και θα συνεχίσουμε τις διαπραγματεύσεις. Δεν είναι κάτι το εύκολο, ιδιαίτερα με την Γενική Διεύθυνση Εμπορίου, αλλά δεν έχουμε επιλογή, είμαστε τέρι, πρέπει να συνεχίσουμε. Τώρα, ως προς το ζήτημα του DCFTA για να σας μιλήσω για το ισοζύγιο πληρωμών. Αρχικά στόχος ήταν να βοηθηθεί η Ορδανία, αλλά τώρα μπορώ να πω ότι η Ορδανία εξάγει στην Ευρωπαϊκή Ένωση 200 εκατομμύρια, ενώ ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση στην Ιορδανία 4 δις. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι γιατί δεν έχουμε φτάσει σε συμφωνίες. Αναφερθήκατε στους πρόσφυγες που έχουν παραμείνει. Η αυτού μεγαλειώτης ε, ζήτησε από την κυβέρνηση να κρατήσει τα σύνορά μας ανοιχτά και τώρα έχουμε πάνω από 2 εκατομμύρια Σύρους, Ιρακινούς, Γεζίντι και ούτω καθεξής. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι έχουμε να κάνουμε με ένα θέμα ασφάλειας που διέπει τον έλεγχο του καθενός που έχει παραμείνει στο έδαφος μας, γιατί προέρχονται και από περιοχές που ελέγχει η ΝΤΑΕΣ. Έχουμε δεχτεί απειλές ότι στέλνουν πυρήνες στην Ιορδανία και μπορεί να προχωρήσουν σε βίες πράξεις. Ελπίζω να να ξέρετε το, το σχέδιο στην Ιορδανία την ε, προηγούμενη εβδομάδα, στη Βόρεια Ιορδανία, εκεί που υπάρχουν περισσότεροι Σύροι, οι δυνάμεις ασφαλείας αντιμετώπισαν έναν μεγάλο τρομοκρατικό πυρήνα συνελήφθησαν περισσότεροι από 30, ορισμένοι σκοτώθηκαν και από τις δικές μας δυνάμεις ασφαλείας και θα ήθελα να πω ότι δυστυχώς υπάρχουν διασυνδέσεις με πρόσωπα από εκείνη την περιοχή. Γι' αυτό έχουμε και ένα θέμα ασφαλείας. Ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχόμαστε ότι καλύτερο κλείνει η συνεδρίασή μας και θα τα πούμε στις 3. Σας ευχαριστώ.